ποιητικά. Και νομίζω ότι έχετε διασώσει την αξιοπιστία, το κύρος και έχετε δείξει την αλληλεγγύη ε, που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις όπως αυτές που μας σχολιάσετε, παραδείγματο χάρη τη Λιβύα. Αυτά που είπατε πράγματι ε, ε, μας κάνουν υπερήφανους ότι έχουμε τριπλάσια βοήθεια σε σχέση με αυτή που παρέχουν είπα για παράδειγμα. Θα ήθελα να σας θέσω τρία ερωτήματα. Μιλήσατε για το συντονισμό στο πλαίσιο της δικής σας εργασίας ε, ε, σε σχέση και με την ΕΙΕΔΑ. Απόψε ο Επιτρόπος Φίλε θα μας παρουσιάσει τη νέα ανακοίνωση για την ανανομένη πολιτική γειτονία. Ένα από τα συστατικά, τα βασικά αυτής της ανακοίνωσης ελπίζω να Αναφέρεται στι δραστηριότητε, των οποίων είστε εσεί υπεύθυνοι στο Σώμα των Επιτρόπων. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση επίσης είδαμε πω η ανακοίνωση η οποία γκρίθηκε πρόσφατα από την Κομισιόν για τις μεταναστευτικές πολιτικές της Ένωσης έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι η δραστηριότητα, η ευθύνη που έχετε εσείς. Και έχω δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό. Είμαστε στο πλαίσιο τη διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού. Εγκρίναμε στην Επιτροπή μα την ομοδότηση που θα στείλουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών. Και θέλω να σα ρωτήσω, οι ανάγκε οι δικέ σα ποιε είναι σε σχέση με τη διαθέσιμα κονδύλια. Καταλαβαίνω ότι θα υπερβούν κατά πολύ οι ανάγκε στα μέσα, τα οποία θα έχετε στη διάθεσή σα, αλλά είμαστε στη διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού. Θα θέλαμε να μα πείτε πώ μπορούμε να σα βοηθήσουμε στο πλαίσιο της δημοσιονομική διαδικασίας. γνωρίζοντα, βέβαια ότι θα πρέπει να κινηθούμε μέσα στα περιθώρια των εφιστάμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Δεύτερη ερώτηση. Εσεί πώ. Ε, ε, συνεργάζεστε με άλλους διεθνείς φόρους, παραδείγματος χάρη τους οργανισμούς ε, των Ηνωμένων Εθνών, ε, την Διεθνή Οργάνωση για τα μεταναστευτικά θέματα κτλ. Είναι ικανοποιητική συνεργασία. Σας γνωρίζουμε ότι τα κονδύλια που απευθύνει στους διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα ήθελα να μας κάνετε έτσι μια περιγραφή της κατάστασης, έναν απολογισμό, πόσο ικανοποιημένοι είστε από αυτή τη συνεργασία με διεθνείς φορείς και οργανισμούς και ιδιαίτερα να ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Σαλαφράγκα, ο συνάδελφο Γκουαλτιέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και εξ ονόματος των ε, Σοσιαλιστών Δημοκρατών για τη σημερινή σας παρουσία εδώ και για την εργασία σας καθώς και για την ε, ενδιαφέρουσα εισήγησή σας για τη συνεργασία εν γέννη που, που έχετε με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και προσωπικά για την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε για τη δική μου έκθεση. περί της ε, άμυνας και της ε, πολιτικής ασφάλειας μετά τη Λισαβόνα. Προσωπικά θα ήθελα να μιλήσω για τις σχέσεις με την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εγώ εκτίμησα ιδιαίτερα και είναι σημείο των καιρών θα έλεγα αυτής της νέας συνολικής προσέγγισης που με κόπο ε, δημιουργούμε Δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά πολλές φορές αν είναι δική σας μια, μια αντιπροσωπεία της Κομισιόν ή αν είναι της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, ή αν είναι εκείνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία όμω και οι πυλώνε δεν υπάρχουν πλέον. Και άρα οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα διάφορα μέσα για να επιβεβαιωθεί μια ενιαίο, ένα ενιαίο όρεμα, ενιαίες αρχές, ένα ενιαίος στόχος. Εκτιμώ λοιπόν αυτή την ε, οπτική. Έπειτα πιο συγκεκριμένα η συγχώνευση αυτών των ε, πυλώνων είναι πολύ πιο περίπλοκη. Και γι' αυτό θα ήθελα να καταλάβω κάπως πιο εις βάθος δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά αυτό το οποίο αναφέρατε, διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε πέρα, εκτός μάλλον της εξωτερικής υπηρεσίας και αυτό είναι κατανοητό. Είναι μάλιστα κοινοτική αρμοδιότητα, υπάρχει διεύθυνση, γενική διεύθυνση. Δεν έχει αυτό ενσωματωθεί στην ΑΕΔ. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Από την άποψη τώρα της ανταπόκρισης της κρίσης, οι οποίες πολύ συχνά είναι κρίσεις όπου εμπλέκονται διάφορες συνιστώσεις. Είναι δύσκολο δηλαδή να ξεχωρίσουμε το τι έχει προκαλέσει ο άνθρωπο, τι όχι, τι έχει πολιτικό αντίκτυπο. Πολύ συχνά μάλιστα μια κρίση γεννιέται λόγω μιας φυσικής καταστροφής, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ασφάλειας. Είναι πολύ περίπλοκες οι καταστάσεις λοιπόν. Συγκεκριμένα λοιπόν πώς μια δομή, ένας φορέας ανταπόκρισης της κρίσης μέσα στην ε, Κομισιόν και το συμβούλια διαχείρισης της κρίσης, κρίσεων μάλλον μέσα στην ΕΙΕΔ θα συνυπάρξουν. Στην ουσία θα έχουμε δύο διαφορετικές δομές που θα συνεπάρξουν. Μία στην υπηρεσία της Επιτροπής και μία στην ε, ΕΕΔ είναι πιθανό να φτάσουμε σε μια συγχώνευση των δύο δομών και μια προφύλαξη των διαφόρων ε, μορφών και νομικών βάσεων των παρεμβάσεων. Δηλαδή η ίδια δομή να είναι στην υπηρεσία δηλαδή της Κομισιόν όταν ε, η αρμοδιότητα είναι κοινοτική και στην και ΕΠΑ όταν είναι απόφαση και αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Θα μπορούσαν δηλαδή να συνεπάρξουν και νομικές βάσεις διαφορετικές που όμως θα διέπουν μια ενιαία υποδομή, μια ενιαία υποδο... Ε, υπηρεσία που θα μπορεί να εξυπηρετεί τα διάφορα θεσμικά όργανα. Ούτως ή άλλως η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν είναι θεσμικό όργανο της ε, Κομισιόν. Την υπηρεσία εξωτερικής δράσης την ε, έχουμε φτιάξει ως μια δομή που εξυπηρετεί όλα τα θεσμικά όργανα, δηλαδή και την Κομισιόν. Απτά. Πρόεδρος. Βάγγελ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε στην Επιτροπή μας. Είμαι ευγνώμων που με τόσο δραστήριο τρόπο ασχολείστε με το έργο σας αυτό. Πιστεύω ότι βάλατε και την προσωπική σας φραγίδα στην επίλυση της κρίσης αυτής και ειλικρινά από τότε που αναλάβατε τη θέση του, της Επιτρόπου ε, κάνατε εξαιρετική δουλειά. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή σαφώς υποδηλώνει ότι υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ αριθμού καταστροφών, αριθμού προβλημάτων τα οποία χειρίζεστε και της αύξησης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός. Αυτή η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό Εξαρτάται επίσης από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί, πολλοί δραστήριοι επίτροποι τώρα που προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Όποτε μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν, με τον ένα ή άλλο τρόπο ασχολούμεθα και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντίδρασης στις ε, κατεπίγουσες ανάγκες. Πολύ συμφωνώ με την ιδέα σας να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο ώστε να λειτουργεί αυτό το θεσμικό όργανο. Αν υπάρχει ένα κέντρο τέτοιο θα είμαστε αποτελεσματικότεροι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πιο αποτελεσματική ως Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μία ερώτηση έχω να σας κάνω συγκεκριμένα. Πώς αλληλεπιδρούν ο πολιτικός και στρατιωτικός τομέας. Στη Σλοβενία γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση τώρα για την πιο δραστήρια συμμετοχή της Σλοβενίας στις επεμβάσεις μετά από κρίση για να σωθούν οι ζωές ανθρώπων που φεύγουν από την Αφρική και πάνε σε χώρες της Ευρώπης. Πολλοί χάνουν τη ζωή τους με τρόπο τραγικό καθοδόν προς την Ευρώπη. Ε, έχουμε ε, σκάφη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες πολιτικές αποστολές. Καταρχήν η κυβέρνησή μας είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους ε, ε, ανθρωπιστικές επεμβάσεις. Εσείς πιστεύετε ότι πρώτον υπάρχει τέτοια ανάγκη, δεύτερον υπάρχει τέτοια δυνατότητα και τρίτον υπάρχει και ένα νομικό θεσμικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να συμμετάσχουμε με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Αν όχι, θα, σας ζητούσα να συνεργαστείτε με άλλους επιτρόπους και με την Επιτροπή συνολικά, ώστε από κοινού να προδιαγράψετε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στα πολιτικά, ε, στις πολιτικές ε, επιχειρήσεις για λόγους ανθρωπιστικούς. Η Επίτροπος θα απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. να απαντήσω στον κύριο Σαλαφράνκα. Δύο θέματα έθιξε. Πρώτον, συντονισμός με την ΕΙΕΔ και άλλους επιτρόπους, όπως τον Επίτροπο Φούλε, τον κύριο Επίτροπο Πίμπαλξ, για τη, μετα, την Επίτροπο Μάλμστρομ για την πολιτική μετανάστευση. Εμείς ε, συνεργαστήκαμε ιδιαίτερα για να εντοπίσουμε τους τομείς που είναι σημαντικοί για την σωστή αντίδραση σε καταστροφές και κρίσεις. Χαρτογραφήσαμε όλες τις περιοχές ε, για να δούμε τους τομείς εργασίας της Κομισιόν και εντοπίσαμε 25 από 26 ε, στους οποίους υπάρχει ένας βαθμός αλληλεπίδρασης. Ποιος δεν μετέχει δηλαδή. Ο Επίτροπος ε, Αλμονία που είναι υπεύθυνο για τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι ο μόνος τομέας που δεν, όπου δεν διαπιστώσαμε αλληλεπίδραση. Γιατί αν δείτε ας πούμε την πρόληψη, την εκπαίδευση, τις υποδομές εκεί, ε, όλα αυτά έχουν γίνει Όσοι προερχόμεθα από σοσιαλιστικό κομμουνιστικό στρατόπεδο ξέρουμε ότι όλοι οι νήσοι κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Η εξωτερική δράση λοιπόν, η αναπτυξιακή συνεργασία, τα... οι εσωτερικές υποθέσεις, αυτά είναι τα... οι τρεις τομείς όπου είχαμε μεγάλη συνεργασία, εντοπίσαμε προτεραιότητες και εντοπίσαμε σε ποια σημεία από κοινού μπορούμε να ε, επιτύχουμε πρόοδο και να υπάρξει κάποια βελτίωση. Βέβαια η δουλειά αυτή ε, εξελίσσεται, αλλά έγιναν πρόοδοι εκεί που χρειάστηκε. Για παράδειγμα με την Επίτροπο Μάλμστρομ συνεργαστήκαμε στενά και για την κρίση στη Λιβύη και για να εντοπίσουμε γενικότερα πώς θα συνεργαστούμε, πώς δηλαδή το νέο κέντρο αντίδρασης στα κατεπήγοντα μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση τρομοκρατικού πλήγματος για παράδειγμα. Κάναμε πρόοδους, αλλά αυτή την ερώτησή σας εγώ την εκλαμβάνω ως ενθάρρυνση για να γίνουν περισσότερα. Τώρα, για τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, ναι, 40% των δραστηριοτήτων μας υλοποιούνται από αυτές τις υπηρεσίες η ΟΤΣΑ, η UN είναι ο πιο σημαντικός εταίρος, ε, τη στηρίζουμε πολιτικά και οικονομικά τη UN και πήγα μάλιστα στα κατεχόμενα και στο Ισραήλ επίσης μαζί με τον Βαλεριάμος, ως ε, ένδειξη ότι συνεργαζόμεθα στην κρίση για τη Λιβύη ε, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες είναι υπεύθυνοι για να πάνε ε, να βοηθηθούν να μεταφερθούν οι πληγέντες. Ε, πολλά πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα στην ανθρωπιστική αντίδραση. Εκεί που εγώ επέμεινα πολύ είναι να φροντίσουμε να είμαστε επικοδομητικοί. Συνεργαζόμαστε μαζί τους ώστε η διαχείριση της κρίσης ε, να υπησέλθει σε σύνθετα θέματα και μετά από μεγάλες καταστροφές. Να έχουμε καλύτερης ποιότητας, δηλαδή προτάσεις. Τι θα κάνουμε δηλαδή συγκεκριμένα. Θα έχουμε ε, ικανότητες διαχείρισης σε εφεδρεία που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται επί 24 ώρου βάσεως ε, κατεπήγοντα. Στη Λιβύη τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά την αντίδραση και στην κρίση του Ιράκ. Είναι δύσκολο το προσωπικό από τα Ηνωμένα Έθνη να μπορεί να έχει την απαραίτητη ε, άδεια εισόδου και κυκλοφορίας. Πρέπει λοιπόν να, εργαστούμε με συντονισμό για να μην λείψουν πρόσωπα. Θα πρέπει όμως να ε, βοηθήσουμε, να επικουρήσουμε την ότσα τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί είναι παράλογο αν εκείνοι δεν παρευρίσκονται στον τόπο όπου χρειάζονται και είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αυτή είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται. Για τον προϋπολογισμό, απευθύναμε έκκληση για να γίνει ε, σεβαστό το ποσό του ενός δι στον προϋπολογισμό ως ελάχιστο απαιτούμενο για να γίνει η δουλειά μας. Αυτό είναι αντιοδικημενικό, στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία. Πέρσι δώσαμε 1,1, δαπανίσαμε 1,1 δις. Στη Παγκόσμια Τράπεζα που την ξέρω, υπάρχει ένας, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας βασικός προϋπολογισμός, ο οποίος δαπανάται κάθε χρόνο. Αν γίνεται αυτό, γιατί πρέπει να προσφεύγω στο αποθεματικό και να μην βάλω τα ποσά που χρειάζομαι στο βασικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν αυτή την ανάγκη. Ο βασικός μας προϋπολογισμός, για λόγους σύγκρισης το λέω, είναι 850 εκατομμύρια. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα χρειαστεί να προσφύγουμε στο αποθεματικό. Ήδη έχει γίνει αυτό. Επίσης, ε, επιμένουμε ότι το αποθεματικό για τις κατεπίγουσες ανάγκες θα πρέπει να είναι ε, διασφαλισμένο. Και θα πρέπει και να αυξηθεί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα φέρει το μέλλον. Το καλό με τα αποθεματικά είναι ότι αν δεν τα, αν δεν χρειαστούμε δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ κάνω χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Όταν θα έρθω του χρόνου σε εσά με προτάσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφών και πώς ε, θα μπορέσουμε το ενεργητικό μας να το ε, αντιστοιχίσουμε με τις ανάγκες. Θα είναι συνετή πρόταση, χρηστή, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε επαρκείς πόρους για να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Κύριε Γκουαλτιέρη, κάνατε πολύ καλή ερώτηση για το αν δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο διαχείρισης κρίσεων που θα καλύπτει τους πάντες. Εγώ επισκέφθηκα τα κράτη-μέλη μας, επισκέφθηκα και κάποιες μεγάλες χώρες, βλέπε η παρουσία την περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί για να δω εκείνη πώς είναι οργανωμένη. Και η προσέγγιση που φαίνεται να είναι η καλύτερη είναι να υπάρχει ένα κέντρο κρίσεων για την προστασία του πληθυσμού των αμάχων για, ε, ως πρώτη αντίδραση και μετά να υπάρχει και το Κέντρο Διαχείρισης Πολιτικών Κρίσεων. Πρόσφατα, ας πούμε, είδαμε τον πρόεδρο Ομπάμα στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, στο Λευκό Οίκο φαντάζομαι θα ήταν αυτό, αλλά υπάρχει πολύ καλά εξοπλισμένη υποδομή στην φήμα που είναι δηλαδή το Federal Emergency Response Agency και ο πρόεδρος ο Ομπάμα ήταν εκεί, τον είδαμε δηλαδή στην οθόνη, στην φήμα, αν πρόκειται για ε, φυσική καταστροφή χωρίς πολιτικο-στρατιωτικές πτυχές. Θα πρέπει οι εντολές να είναι διακριτές και η ανθρωπιστική ανάγκη η προστασία των αμάχων, η πολιτική προστασία έχει συγκεκριμένους στόχους. Βέβαια, ε, στην περίπτωση των ΙΠΑ, ο επικεφαλής των ΦΥΜΑ μπορεί να κληθεί να καθίσει στο κέντρο όπου ε, θα γίνεται η πολιτικοστρατιωτική διαχείριση της κρίσης. Και εμείς προς τα εκεί κινούμεθα. Στην Ευρώπη εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, σημαντικό. Οι υπηρεσίες μου είναι υπεύθυνε για να αντιδρούν στις καταστροφές και μέσα στην Ευρώπη. Πλημμύρες ή κόκκινη λάσπη πέρσι ή τώρα με το πρόβλημα του ηφαιστείου ελπίζω να ηρεμήσει σύντομα, αλλά αν πει η Ισλανδία πρέπει να μας βοηθήσετε, πρέπει να πάμε και να αναπτύξουμε δυνάμεις εκεί και έτσι είναι δύσκολο αυτό να συμπεριληφθεί στην ΕΕΔ. Ε, Αλλά στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη ΣΥΠΑ είδα ότι για τα ανθρωπιστικά και τις φυσικές καταστροφές υπάρχει ένα ειδικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων που συνδέεται με το κέντρο πολιτικής προστασίας Εκεί που πρέπει να δουλέψουμε όμως είναι στον εξή τομέα και πάω στο, στη δεύτερη ερώτηση. Να εντάξουμε άλλες ε, κρίσεις επισητιστικές, κρίσεις ασφάλειας ε, όταν είχαμε την ε, συγκεκριμένες επιδημίες. Τι θα γίνει αν προκύψει ξαφνικά μια οξία κρίση. Θα πρέπει να προβλέπετε η αντιμετώπιση. Να έχουμε δηλαδή μικρά κέντρα αντιμετώπισης επιμέρους κρίσεων. Και θα πρέπει να συζητήσουμε αν μπορούμε όλα αυτά να τα εντάξουμε σε ένα κέντρο ενιαίο στην Κομισιόν. Και αν έχουμε περισσότερα κέντρα, εντάξει, αλλά πρέπει να είμαστε ορθολογικοί. Να κάνουμε μία ανάλυση. Αυτό το συζητήσαμε και με τον Αντιπρόεδρο Σευκόβι και προχωρούμε σε μια αντικειμενική αξιολόγηση για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Κυρία Βάιγκελ, εκτιμώ το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι λένε ότι πρέπει να είμαστε ε, ε, τμήμα μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής, ε, στον κύριο Βάγκελ, προσέγγισης. Και αυτό σκέπτεστε και στη Σλοβενία. Τώρα, αν κάποιο σκάφος ε, του στόλου σας μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των ε, προβλημάτων που έχουμε με τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη. Καταρχήν, αν υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει, είναι η Frontex. Ο ρόλος της Frontex ε, είναι μετά από αίτημα των κρατών μελών να παράσχουν βοήθεια και στον τομέα της ασφάλειας, αλλά να σώζουν και ζωές εάν αυτό χρειαστεί. Αυτή, ε, η βοήθεια γίνεται μετά από αίτημα κράτους που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Η Ιταλία εν προκειμένου. Αν το ζητήσει η Ιταλία μπορεί τότε αυτό το σκάφος του στόλου σας να ενταχθεί στις επιχειρήσεις της Frontex. Για μας, για την ανθρωπιστική κοινότητα, εμείς χρησιμοποιούμε ε, υποδομή των ενόπλων δυνάμεων για να ε, αντιμετωπίσουμε πολιτικά προβλήματα, όπως το Πακιστάν για παράδειγμα, όπου ε, στείλαμε τα, τη βοήθεια με στρατιωτικά σκάφη, στη Λιβύη για την εκένωση περιοχών ή απομάκρυνση υπηκών τρίτων χωρών. Το κρίσιμο θέμα είναι όλα αυτά να είναι υπό την αιγίδα του πολιτικού ελέγχου, ούτω ώστε να μην στρατιωτικοποιούμε μια ανθρωπιστική επιχείρηση. Θέλω να τιμήσω το στρατιωτικό προσωπικό της Ένωσης, γιατί έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί τους. Η στρατιωτική ηγεσία μας επέτρεψε να διαμορφώσουμε σαφές ξεκάθαρο πρωτόκολλο και καμιά φορά οι αξιωματική τους ε, έπαιξαν το ρόλο των αξιωματικών συνδέσμων στις δικές μας δυνάμεις ε, διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν μπορούσαμε να εντάξουμε κράτη-μέλη σε αυτή τη συντονισμένη αντίδραση η οποία σημαίνει ότι θα σώσουμε περισσότερες ζωές και θα παράσχουμε περισσότερη βοήθεια. Ευχαριστώ. Επόμενη σειρά ερωτήσεων με τον συνάδελφο Κιλ Νίλσεν των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας παρουσίαση και να σας συγχαρώ διότι διοριστήκατε, ε, μάλλον ε, εκλεγήκατε, επίτροπος ε, της χρονιάς. Σας συγχαίρω και εκφράζω την χαρά μου γι' αυτό. Εμεί εκφράσαμε τη λύπη μα ότι δεν υπήρχε αρκετά πολιτικό προσωπικό για τι ε, αποστολέ πολιτικού τύπου. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να βελτιώσετε την κατάσταση. Επίση είπατε ότι μεταβήκατε στα Παλαιστινιακά εδάφη, ε, επισκεφθήκατε το Σεξαρά, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου είδατε οικογένειε που διαρκώ ε, διώκονται από τι κατοικίε του Βεδουίνου Παλαιστινίου είδατε επίση που επίση διώκονται από τα χωριά του και τα σπίτια του. Μιλήσατε για τη Γάζα όπου σίγουρα θα συμφωνήσετε ότι δεν βρισκόμαστε ενώπιον μια φυσικής καταστροφής αλλά ενός ε, πολιτικού προβλήματος και ε, μου έμεινε μια φράση που πάτε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να είναι πολιτικό εργαλείο. Διερωτώ με λοιπόν σε σχέση με το μπλοκάρισμα το, το εμπάργο της ε, Γάζας. Ε, είναι ένα παράνομο εμπάργο που οδηγεί σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση. Πριν από αυτό, οι 10% των κατοίκων της Γάζας εξαρτώνταν από την ανθρωπιστική βοήθεια και τώρα έχουν φτάσει στο 70 με 80%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει, πληρώνει το ποσό που αφιερώνεται στην ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστινίους και μάλιστα και στις, ε, στα διάφορα στρατόπεδα προσφύγων ε, πληρώνει πολλά χρήματα και αν δεν θέλουμε να συνεχίζουμε να τραβάμε από τα αποθυματικά μας όπως είπατε θα πρέπει να βρεθεί πολιτική απάντηση σε αυτή την κατάσταση που δεν πρέπει πια να κρατήσει άλλο. Πρόκειται σαφώς για πολιτικό πρόβλημα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ανθρωπιστική απάντηση. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να προχωρήσουμε λοιπόν για το θέμα αυτό και να μην αρκούμεθα Λυπάμαι που το λέω έτσι άμεσα. Εσείς είπατε ότι παρακαλέσατε το Ισραήλ, το εκλυπαρίσατε μάλιστα, ε, για να σταματήσει το εμπάργο. Μα δεν αρκεί αυτό όμως, δεν ακούν τα παρακάλια. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο σταθεροί και αυστηροί απέναντι σε αυτό το παράνομο ε, εμπάργο. Να υπογραμμίσω κάτι ακόμα που νομίζω να είναι σχετικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή χάνει την αξιοπιστία τη απέναντι στου Ευρωπαίου πολίτε για αυτό ακριβώ το ζήτημα. Και νομίζω πω η παράλυση, η πολιτική παράλυση τη Ένωση απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ε, όλο ένα και λιγότερο γίνεται κατανοητή και όλο ένα και λιγότερο είναι αποδεικτή από του Ευρωπαίου πολίτε. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπω και εγώ, ότι ένας νέος τολίσκος είναι έτοιμος να φύγει για τη Γάζα, 15 σκάφη τα οποία έχουν αυλώσει πολίτες μη βίαιοι που επιθυμούν ακόμα μια φορά να καταγγείλουν το παράνομο εμπάργο της ε, λωρίδας της Γάζας και να απαιτήσουν γρήγορα δράση για να σταματήσει αυτή η κατάσταση που διαρκώ επιδεινώνεται. Άκουσα την κυρία Άστο να λέει πως δεν ήταν καλή απάντηση. Ίσως, αλλά οι πολίτες οι πολίτες προσπαθούν ανθρώπινα να απαντήσουν με μη βίαιο τρόπο σε μια κατάσταση που είναι πια αναβάσταχτη. Εγώ προσωπικά έχω επισκεφθεί πολλές φορές την Γάζα τους τελευταίους μήνες και πρέπει να σας πω ότι κάθε μου επίσκεψη είναι και πιο αβάσταχτη. Γιατί βλέπουμε την κατάσταση διαρκώς να επιδεινώνεται. Η ερώτησή μου είναι η εξή και η κυρία Άστον είπε ότι ο στολίσκο δεν είναι λύση και σε αυτό το στολίσκο θα είναι μη βίαιοι πολίτε. Θα υπάρχουν και τοπικοί και περιφερειακοί αλλά και ευρωβουλευτέ. Ε, ε, ε Πολύ και διάφοροι λοιπόν. Τι προτίθεστε να κάνετε για να προστατεύσετε τους Ευρωπαίους πολίτες και να μην υπάρξει νέο δράμα όπως πέρσι με το πρώτο στολίσκο. Σας ευχαριστώ. Bene, l'onorevole Galler è il prossimo a intervenire. Ja, vielen Dank. Vielleicht gleich eine Reaktion auf die Vorrednerin. Ich bin davon überzeugt, dass ich... Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα πρέπει να υπάρξει, να υπάρξει μια πολιτική δράση, ε, αλλά δεν θέλω να προδικάσω τις απαντήσεις της Επιτρόπου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το... την αφοσίωση με την οποία ασχολείστε με τα καθήκοντά σας. Βλέπω ότι έχετε σαφή προσανατολισμό και θέλετε μια γενική διεύθυνση η οποία θα διέπεται από ε, συγκεκριμένες πολιτικές ώστε και οι υπάλληλοι να ξέρουν ε, τι γραμμή πλεύσης θα ακολουθήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε γιατί καμιά φορά αναρωτιόμαστε ποια είναι η προστιθέμενη αξία άλλων πολιτικών. Ε, συγχαρητήρια λοιπόν καταρχήν. Μια γενική ερώτηση σχετικά με τα διάφορα μέσα που διαθέτουμε. Έχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Λειτουργεί. Πάει καλά πιο μακροπρόθεσμα, έχουμε το DHI και μακροπρόθεσμα και αναπτυξιακή βοήθεια για την ε, ανοικοδόμηση. Αλλά το πρόβλημα είναι, νομίζω, εδώ, ότι η Κομισιόν δεν ε, χρησιμοποιεί έγκαιρα τα μέσα που διαθέτει μετά από μια ανθρωπιστική κρίση. Είναι λίγο δυσκίνητα τα προγράμματα. Παίρνει ένα-δύο χρόνια μέχρι να λειτουργήσουν απόλυτα. Και χρησιμοποιείται το μέσο σταθερότητα επειδή είναι πιο εύχριστο αλλά δεν είναι πρικοδοτημένο επαρκώς. Όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα και δυνατότητες επέμβασης ε, συζητούνται από την Επιτροπή, από όλους τους επιτρόπους ή θα θέλατε να δώσετε εσείς το έναυσμα για μια σχετική συζήτηση ούτως ώστε να ε, υπάρχει έγκαιρη δράση με επαρκή κονδύλια. Αυτή είναι μια γενική ερώτηση. Τώρα για τη Λιβύη συγκεκριμένα είπατε ότι η U4 είναι έτοιμη αλλά επεμβαίνει μόνο όταν η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι εγγυημένη. Αυτό είναι σαφές. Και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την ΟΤΣΑ. Ή μάλλον η ΟΤΣΑ μόνη της αποφασίζει. Πιστεύετε ότι ε, η ότσα συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ελεύθερη από πολιτικές επιρροές. Ρωσία-Κίνα που ενδεχομένως θα έβαζαν βέτο. Η διαπίστωση δηλαδή ότι η ανθρωπιστική ε, πρόσβαση δεν είναι διασφαλισμένη, αυτή η απόφαση λαμβάνεται ή μπορεί να λαμβάνεται μόνο από την Ότσα ή θα πρέπει και εμείς να ε, αποφασίσουμε αν δεν γίνεται ή αν δεν μπορεί να αποφασίσει η ότσα, τότε θα μπορούσε και χωρίς την ότσα να ε, χρησιμοποιηθεί η u 4 Ευχαριστώ. Είναι τώρα η σειρά του συναδέλφου Κυρίλοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, με εντυπωσίασε η ενδιαφέρουσα σας παρουσίαση και τεράστιες προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε και κάποιες φορές ε, ε χωρίς να έχετε προετοιμαστεί γι' αυτό και για την ώρα ε, δίνετε τις κατάλληλες απαντήσεις. Ε, έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, η μία σε σχέση με αυτή του προηγούμενου συναδέλφου για τη Λιβύη. Φυσικά δεν εξετάζω τις ε, υποχρεώσει εξωτερικής πολιτικής, αλλά όσον αφορά την πρόσβαση στους ε, πολιορκημένους ανθρώπους διαφόρων κοινοτήτων ε, δυτικά της Τρίπολης στην Ιεφρέν, που ήδη κάνουν δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια τους τελευταίους δύο μήνες. Προφανώς η υπόθεση της Λιβύης είναι πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά την στρατιωτική και πολιτική συνεργασία. Εφόσον δεν μπορούμε να βάλουμε πόδι λοιπόν επί τόπου, μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες να στείλετε βοήθεια από αέρο στις πιο στις, στις, στις ε, καταστάσεις όπου τους λείπουν τα πάντα, τρόφιμα, ε, φάρμακα και ούτω καθεξής. Τώρα κάτι άλλο κάθε φορά που συμβαίνει. Τώρα, ακριβώ πριν από το καλοκαίρι, μπορούμε με ασφάλεια να προγραμματίσουμε, τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουμε όμω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για του πολίτε μα, να δουν δηλαδή την αλληλεγγύη, την ευρωπαϊκή δράση μέσα στα σύνορά μα. μπορούμε να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι και ενεργούμε κοινά. Συμβαίνει συχνά Για τις πυρκαγιές η Ελλάδα ζητούσε βοήθεια από τη Ρωσία για τούμπαλ είναι ας πούμε. Ε, είναι πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε questions uh, uh, uh, Ευχαριστώ. Καταρχήν, το ευρύτερο θέμα. Αν έχουμε δηλαδή πολιτικό-στρατιωτικό δόγμα ή μοντέλο λειτουργίας. Ναι, είναι η απάντηση. Έχουμε και στηρίζεται σε, τρεις, σε τρία μέρη. Πρώτον, τα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν επί κατευθυντηρίων γραμμών για το πώς θα λαμβάνει η χώρα η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία και εμείς δεσμευόμεθα ως Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές που ε, ορίζουν πώς θα χρησιμοποιηθεί το στρατό, σε έσχατη λύση κλπ. Ορίζεται ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να γίνεται με πολιτική εποπτεία. Και αυτό γιατί, γιατί θέλουμε πάντοτε να εξαντλούμε κάθε πιθανό τρόπο, κάθε δυνατότητα να φτάσουμε σε κόσμο που είναι ουδέτερος. Γιατί αυτό προστατεύει τη ζωή των ε, εργαζόμενων στην ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα στον κόσμο. Πέρυσι, περισσότεροι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια πέθαναν από ότι αυτοί που συμμετείχαν σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Και φέτος πιθανότατα θα γίνει το ίδιο αλλά είναι και απαραίτητη η δουλειά αυτή, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, θέτουμε, δημιουργούμε φρικτά παραδείγματα που μπορεί να τα εκμεταλλευτούν οι διάφορες. Σκεφτείτε το Σουδάν και την Δημοκρατία του Κονγκό και ένα σωρό με παράξενα μέρη όπου γίνεται χαμός και αν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις κατευθύνες γραμμές φυσικά δεν εξυπηρετούμε τίποτα. Άρα λοιπόν, ε, ναι, ε, στρατιωτικές ε, και αμυντικές δυνάμεις στι ανθρωπιστικές αυτές αποστολές. Λοιπόν, έχουμε και τις, το ανθρωπιστικό κομμάτι και τα προηγούμενα που δημιουργήσαμε στο παρελθόν και που δείχνουν πώς εφαρμόζουμε το, την αρχή της έσχατης λύσης ή καταφυγής και αυτά τα προηγούμενα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για όλους μας, γιατί κάθε περίπτωση διαφέρει βέβαια, αλλά ε, μαθαίνουμε από όλα αυτά. Όταν πήγα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, όταν πήγα στο Ισραήλ ως επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια, πήγα για να ενισχύσω τη φωνή των πιο ευάλωτων ανθρώπων που ήταν το 62% της δυτικής ε, όχθης υποκατοχήν από το Ισραήλ, αραιοκατοικημένη περιοχή, κυρίως ε, βεδουίνων φυλές ε, είναι εκεί και είχα την δυνατότητα να προβάλλω το αίτημά του στο βασικό. Δηλαδή λένε παρακαλώ επιτρέψτε μας ε, να προχωρήσουμε τα αιτήματά μας για δόμηση κλπ. Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, οικογένειε ηλικιωμένων που ε, έγινε έξωση από τα σπίτια και στη Γάζα δυστυχώς επιδεινώθηκε η κατάσταση. Η, ε, βοήθησε λίγο η πολιτική του Ισραήλ από τον προηγούμενο Ιούνιο που χαλάρωσε τα μέτρα και έρχονται πιο πολλά καταναλωτικά αγαθά και τρόφιμα στη Γάζα, αλλά της διπλής χρήση είναι πολύ περιορισμένα, οπότε η οικονομική δραστηριότητα δεν τονώνεται αν υπάρξει πρόσβαση στη Γάζα δεν υπάρχει πρόβλημα ανθρωπιστικής βοήθειας. Η λύση είναι πολιτική βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι η δική μου δουλειά. Η δική μου δουλειά είναι να φροντίσω ότι η βοήθεια θα, ε, θα είναι καλά στοχευμένη για ε, προστασία των πιο ευάλωτων, νομικές συμβουλές, βοήθεια στους ανθρώπους που τους έγινε έξωση για να μην μείνουν στο δρόμο, τρόφιμα και ψυχολογική υποστήριξη στο πληθυσμό της Γάζας. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικών διαπραγματεύσεων για να υπάρξουν αποτελέσματα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο λαός της Παλαιστίνης και η ηγεσία του θεωρούν ότι το Σεπτέμβριο πρέπει να ε, κάνουν εκλογές. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό. Και η Ισραηλινή ηγεσία, από ό,τι κατάλαβα, ακόμα εξετάζει τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο και τι σημαίνουν αυτές. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα ασφαλείας, επισκέφθηκα ένα χωριό ε, που είναι κοντά στη Γάζα και παίζουν τα παιδιά σε καταφύγια, αφύσικα πράγματα. Δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση ούτε εκεί. Αλλά η δική μου, το δικό μου μέλημα είναι ότι υπάρχουν πολλοί Παλαιστίνοι που υποφέρουν και εγώ τι κάνω, τους αντιμετωπίζω με ε, ασπιρίνες, ενώ η λύση είναι πολιτική. Κύριε Γκάλερ, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αναγνωρίζετε τις καλές υπηρεσίες των συνεργατών μου που είναι εξαιρετικοί. Οι 300 ιδιαίτερα που καλύπτουν όλο τον κόσμο και πάνε στην Ιεμένη, στα κατεχόμενα, στο Σουδάν, στον Ταρφούρ, είναι πολύ γενναίοι άνθρωποι, θαραλέοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες και αξίζουν να υποστηριχθούν στο έργο τους. Εμείς αναγνωρίζομαι ε, ιδιαίτερα και εκτιμούμε το ζήτημα που θέσατε. Μπορεί γρήγορα να γίνει η ανθρωπιστική βοήθεια. Είμαι η μόνη επίτροπος, μπορώ να αποφασίσω σε 24 ώρες και δυστυχώ πρέπει να παίρνω εσπευσμένα αποφάσει συχνά. Συνήθω το έργο μας διαρκεί 6 με 9 μήνες, μάξιμου. Κανένα φορά μένουμε λίγο παραπάνω. Και τα μέσα τα αναπτυξιακά είναι τόσο βραδέα ώστε δημιουργείται ένα κενό με τον Επίτροπο Πίμπαλξ. Είχαμε αποφασίσει δύο προτεραιότητες συνεργασίας για την αναπτυξιακή συνεργασία και την αντιμετώπιση καταστροφών. Τώρα, πάλι με βάση το υπόβαθρό μου από την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι ότι λείπει κάτι, ένα ευέλικτο μέσο που θα καλύπτει το κενό και θα ε, έχει να καλύψει την πρώιμη ανασυγκρότηση και θα μπορούν και οι δύο υπηρεσίε να συνεργάζονται πάνω σε αυτή τη βάση. Ραγίζει η καρδιά μου στον Ταρφούρα που πήγα σε ένα καταβλισμό ε, όπου δίναμε τρόφιμα αλλά δεν δίναμε ελπίδα γιατί τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να ε, προσφέρουμε εκπαίδευση, να δώσουμε τρόφιμα αλλά δεν, δεν εξασφαλίζουμε μια αξιοπρεπή ζωή μακροπρόθεσμα. Και μίλησα και με τον Μπομπ Ζέλικ που ήταν ο πρώην ε, ε, προϊστάμενός μου για αυτό το θέμα. Δεν το συζητεί συχνά. Ε, είπε, όχι δεν χρειάζονται νέα μέσα και μηχανισμοί. Δεν ξέρω ποια είναι εδώ η νομική κουλτούρα μας, αλλά η δικαιική. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος χρηματοδότησης για να βοηθάμε τον κόσμο. Αλλιώς συνεχώς θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο όταν ε, είναι έτοιμη η ανθρωπιστική βοήθεια αλλά όχι η αναπτυξιακή συνιστόσα. Τώρα έχουμε εντοπίσει περιπτώσεις όπου με τον Επίτροπο Πίμπαλξ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια διαφορά. Ας πούμε στην ακτή του ελεφαντοστού έχουμε σημαντική ε, βοήθεια ανθρωπιστική 60 εκατομμύρια, εκείνος έχει 180 εκατομμύρια ε, αναπτυξιακή συνεργασία και προσπαθούμε να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση ευθύς εξ αρχής. Και θα έρθω να σας πω ε, τι θα γίνει από εκεί ε, και αν πετύχαμε. Ο κύριος Κύριλοφ. Για μισό λεπτό τώρα γιατί... Α, ε, θυμάμαι, δύο ερωτήσεις κάνατε. Μία για την Ότσα. Αν η Ότσα όχι, αυτό ήταν η ερώτηση του κυρίου Γκάλερ για την Ότσα και τη u Ναι, ναι, ναι, με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα λιγάκι με τις ερωτήσεις και τη, τους ερωτώντες. Για την Ότσα και τη u Υπάρχει ανθρωπιστική πρόσβαση ακόμα, δύσκολη, με πολλούς περιορισμούς, αλλά υπάρχει ακόμα. Η Ότσα προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια ανθρωπιστική προσέγγιση που θα επιτρέπει την παροχή της ε, ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Θα δούμε αν θα πετύχει. Υπάρχει λοιπόν πρόσβαση, ελπίζουμε να ε, διευρυνθεί, πρέπει να το πιέσουμε αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι γίνει αν στα πλαίσια της παρούσας εντολής η Ότσα καλέσει την U4. Αυτή η εντολή περιορίζεται σε μια επιτόπια βοήθεια. Τι παραπάνω μπορεί να κάνει κανείς αυτό που δεν μπορεί να κάνει τώρα το ΝΑΤΟ. Πώς ας πούμε τα παραδοτέα τους θα είναι περισσότερα. Αν τα Ηνωμένα Έθνη δεν αλλάξουν το ψήφισμα που είναι απίθανο για να επιτραπεί η παρουσία της, η U4 νομίζω ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά εμπόδια. Ναι, είναι καλό να υπάρχει μια ακόμα εναλλακτική, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούν να κάνουν αυτοί. Αλλά το καλύτερο είναι να πιέσουμε για ανθρωπιστική πρόσβαση. Ε, τώρα, στην ερώτηση του κυρίου Κύριλοφ. Μέχρι τώρα δεν ζητήσαμε από το ΝΑΤΟ να κάνει ρήψεις ε, ανθρωπιστικής βοήθειας ε, γιατί στις περιοχές που ελέγχονται από τον Καντάφη ε, δεν ξέρουμε αν πετάξουμε κάτι από πάνω σε ποιανού τα χέρια θα πέσει. Είναι πολύ πιθανό να πέσει βοήθεια στα χέρια του στρατού του Γκαντάφη που θα σπεύσουν πρώτοι επιτόπου. Και αυτό που εξακολουθούμε να βλέπουμε και το λέω ως εμπιστευτικό. Ε, η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις μπόρεσαν να επιτόπου να φτάσουν στον κόσμο. Δεν το διαφημίζουν πάρα πολύ αυτό λόγω θεμάτων και προβλημάτων ασφαλείας. Δεν θέλουν δηλαδή να στρέψουν την προσοχή των δυνάμεων του Καντάφη σε αυτά που κάνουν. Ε, υπάρχει λοιπόν ως ένα βαθμό περιορισμένο αλλά κάποια πρόσβαση εξακολουθούμε να έχουμε. Α, για τις ε, δασικές πυρκαγιές επίσης ρώτησε ο κύριος Κύριλοφ. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γιατί ήταν δική σας πρωτοβουλία να έχουμε φεδρική ικανότητα για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Τώρα θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα από αυτά και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τα κράτη-μέλη μας αύξησαν την ικανότητά τους, αλλά δεν πειράζει να βοηθήσει και η Ρωσία, γιατί η Ρωσία, εις ό,τι αφορά τις ικανότητες καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών, είναι πολύ προχωρημένη. Και ήθελα και με τον ε, ε, Υπουργό Σόιχου να δούμε τι συμφωνίες συνεργασίας μπορούμε να έχουμε. Τώρα, εις ό,τι αφορά την ε, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έχουμε πολλά να κάνουμε. Και κάνω έκκληση εδώ. Υπάρχει ένα ταμείο που λέγεται Ταμείο Αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Ο σκοπό του είναι αν υπάρξει καταστροφή και αν είναι πιο δαπανηρή από το 0,6 του ε, ΑΕΠ να ε, παρέμβει το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ωραία. Αλλά είναι πολύ δυσκίνητο αυτό το Ταμείο και ε, παίρνει αιώνες μέχρι να φτάσουν τα χρήματα. Είχαμε τις πλημμύρες στη Ρουμανία συνεχίστηκαν, μετά έγιναν πλημμύρες στη Μολδαβία. Στη Μολδαβία μέσα σε 24 ώρες μπορώ να τους δώσω μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια. Στη Ρουμανία όμως δεν μπορώ. Δεν είναι παράλογο αυτό. Πρέπει λοιπόν να ανακαινήσουμε αν θέλετε το Ταμείο Αλληλεγγύης για να γίνει ταχύτερο και να μπορούμε να δείχνουμε αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη μας όπως δείχνουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε πολλά να κάνουμε εσωτερικά λοιπόν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν θα περιόριζα την απόκριση στις καταστροφές μόνο στην Ευρώπη. Συζητάμε και με την Αυστραλία και με τη Νέα Ζηλανδία μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Όταν είναι καλοκαίρι εδώ, στους αντίποδες είναι χειμώνα. και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δικές τους ομάδες να μας βοηθήσουν στο δικό μας καλοκαίρι και να στέλνουμε, να, βοηθάμε εμείς όταν έχουν εκείνη καλοκαίρι. Αυτή είναι μια συμφωνία συνεργασίας που συζητάμε. Γιατί σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο απρόβλεπτος από φυσική και πού θα πλήξει η καταστροφή, σε ένα τέτοιο κόσμο πρέπει να έχουμε παγκόσμια συνεργασία. Αυτή είναι μια γενικότερη πρόκληση για την κοινότητα των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος Ζώ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των συναδέλφων για τη σαφήνεια των, των απαντήσεών σας. Όλοι εκτιμήσαμε την εισήγησή σας και τις απαντήσεις που δώσατε πολύ συγκεκριμένες και πολύ εις βάθος. Φυσικά θυμήσατε τις ανθρωπιστικές ε, δράσεις και τις ε, δράσεις βοήθειε για τι φυσικέ καταστροφέ, τι ανθρώπινε καταστροφέ, δεν είναι πολιτικές, δεν θα πρέπει να πολιτικοποιούνται, όμω εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ έντονες πολιτικέ δράσει για του πολίτε μα. Και όπω τόνισαν αρκετοί συνάδελφοι, ο κύριος Αλαφράγκα και ο κύριος Κύριλοφ, ε, σε μια περίοδο όπου σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, πολιτικό, χρηματοπιστωτικό, είναι κάποιε φορέ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορθώσει το ανάστημά τη και να δείξει και να Νομίζω πως το θέμα τα οποία εσείς έχετε αναλάβει είναι μια απάντηση που δίνουμε και στους πολίτες μας να τους δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αλληλεγγύη υπάρχουν και είναι και αποτελεσματικέ και εκεί παίζετε εσείς κυρίαρχο ρόλο. Η ενέργεια και η αποφασιστικότητα που μας δείξατε σήμερα θα θέλαμε εμείς οι βουλευτές να τη βλέπουμε ε, και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας και στο πολιτικό και στο στρατιωτικό επίπεδο δώδαμε συγκεκριμένα στην κρίση της Λιβύης. Ε, συγχαρητήρια λοιπόν για το έργο σας και να έρχεστε να μας βλέπετε πιο συχνά. Ευχαριστώ. Αντίο σας. Colleghi, prima di passare Πριν περάσουμε στο σημείο 12, τον απολογισμό της αποστολής της αντιπροσωπείας ερχόξαν Βανίας 6 και μέχρι 9 Μαΐου από τον Έντορ Κούκαν που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα από τη Βοσνία Ριζεγοβίνη που παρακολουθεί τη συζήτησή μας. Πού βρίσκεστε, χαιρετίστε μας. Καλωσορίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η συνεργασία με τα κοινοβούλια της περιοχής είναι για μας πολιτική προτεραιότητα. Και η δική σας παρουσία εδώ είναι ένα θετικό μήνυμα για το θετικό ενδιαφέρον που έχετε για την Ευρώπη. Σας εύχομαι να διασκεδάσετε με αυτή τη συζήτηση. Να περάσουμε στον απολογισμό της αποστολής αντιπροσωπείας ad hoc στην Αλβανία που έγινε 6 με 9 Μαΐου με τη ευκαιρία των δημοτικών εκλογών που έγιναν στη χώρα. Παρακολουθήσαμε με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης και την αύξηση των πολιτικών εντάσεων στη χώρα. Ε, έγιναν πρόσφατα διαδηλώσεις ε, διαμαρτυρίας ε, στα Τύρανα και ε, γι' αυτό ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο επίτροπος Φίλε αποφάσισαν να αναβάλουν την προβλεπόμενη επίσκεψή τους στη χώρα για αργότερα. Εσείς κύριε Κούκαν με μεγάλη διπλωματικότητα ηγηθήκατε της ε, αντιπροσωπείας μας εκεί και σας δίνω το λόγο για να μας εξηγήσετε τι ε, αντιμετωπίσατε επί τόπου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις διάφορες πολιτικές ομάδες γιατί ενδιαφέρθηκαν για αυτές τις εκλογές και για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής. Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να στείλει μια ad hoc αντιπροσωπεία στην Αλβανία για να παρατηρήσει τις ε, τοπικές εκλογές που έγιναν στις 8 Μαΐου 2011. Ήμασταν ε, μια αποστολή ε, περιορισμένη σύνθεσης ε, και το ακολουθήσαμε την συνηθισμένο, τα συνηθισμένα όσον αφορά την αποστολή. η αποστολή αποτελείται από μένα και άλλους τρεις ε, Ο Γιώργος Κουμουτσάκος από ΕΛΚΑ από την Ελλάδα και ο Μιχαήλ Τρεμόπουλος από τον Πρασίνων ΕΦΕ από την Ελλάδα. Επίσης και τον κύριο Στάινουρκ. Είχαμε επαφέ με την κοινωνία των πολιτών, διεθνεί εκπροσώπου στη χώρα, την παραμονή των εκλογών. Ε, ε, επισκεφθήκαμε αστυνομικού σταθμού, ε, συγγνώμη, ε, εκλογικά κέντρα ε, την ημέρα των εκλογών, αλλά δεν μπορούσαμε να προβούμε σε αξιολόγηση της εκλογικής διαδικασίας του ίδιας και αυτό ε, είναι παράθεση από την επιστολή του Πρόεδρου Μπούζεκ στην ε, Πρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου, κυρία Τουπάλη. Ήρθαμε σε επαφή με διάφορους ηγέτες των κομμάτων, εκπροσώπους της διπλωματικής κοινότητας, τα ΜΜΕ και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ακούσαμε για τις πολιτικές εντάξεις και την πόλωση της εκλογικής εκστρατείας. Η σοσιαλιστική αντιπολίτευση έκανε διάφορους ισχυρισμού όσον αφορά υποτιθέμενες πιέσεις που ασκήθηκαν σε δημόσιους υπάλληλους και ε, ε, περιπτώσεις ε, πλαστοποίησης ταυτότητας είχαμε και άλλα μέρη, παρατηρήσαμε και άλλα εκλογικά κέντρα στην Αλβανία. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εν γέννη η εκλογική διαδικασία ήταν τακτική και ειρηνική. Αυτό ήταν ευπρόσδεκτο από όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας λόγω της πολιτικά απολωμένης κατάστασης της χώρας και την ε, ε, άκρα πολιτικοποίηση της προεκλογικής εκστρατείας. Ορισμένα θέματα που αφορούσαν τη διαδικασία ψηφοφορίας παρατηρήθηκαν από την αντιπροσωπεία και αξίζει να τα αναφέρουμε. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήσαμε οικογενειακή ψήφο. Επίσης είδαμε καθυστερήσεις στο άνοιγμα και σύγχυση στο κλείσιμο των εκλογικών κέντρων μεγάλες μακριές ουρές ε, τόμων παρατηρήθηκαν σε πολλά εκλογικά κέντρα. Επιπλέον η καταμέτρηση είχε κεντροποιηθεί και αυτό δημιουργούσε ερωτήματα για διάφορες κοινότητες και προκάλεσε και κάποιες ερωτήσεις στη διαδικασία καταμέτρησης σε ορισμένου δήμους. Ιδιαίτερα στην ε, πρωτεύουσα στα Τύρανα η καταμέτρηση πήρε πάρα πολύ ε, χρόνο ενώ τα προκαταρτικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 14 Μαΐου. Τελικά ο Έντι Ράμα πήρε τις περισσότερες ψήφους από τους σοσιαλιστές. Διοπιστώσαμε την ημέρα των εκλογών, όπως σας είπα, ότι έγιναν ειρηνικά και τακτικά οι εκλογές. Αρκετές βελτιώσεις έγιναν, σημειώθηκαν συμπεριλαμβανομένων των ε, Ε, παρατηρήσεων ε, αυτών ε, νομίζω πως αυξήθηκε η κυριότητα της εκλογικής διαδικασίας. Όλοι δε οι Αλβανοί συνομιλητές μας καλωσόρισαν ως θετική την παρουσία του Ευρωκοινοβουλίου και ως προς αυτό πιστεύω ότι η παρουσία της διεθνούς κοινότητας και των παρατηρητών της είναι χρήσιμη και ουσιαστική. Μέχρι στιγμή λοιπόν όλα καλά, εμείς εκπληρώσαμε την εντόλη, αλλά λόγω των εξελίξεων στη χώρα μετά από την ημέρα των εκλογών. Νομίζω πως δεν μπορώ να σταθώ στα αυτά. Θα πρέπει να σας ενημερώσω για την κατάσταση. Μετά από την ημέρα των εκλογών αντιμετωπίζουμε μια επιδείνωση της κατάστασης. Υπήρξαν εξελίξεις μετά από τα, πριν από την ανακοίνωση των προκαταρτικών αποτελεσμάτων από πλευράς της ΟΑΣΕ στις 14 Μαΐου ε, η Συμμαχία των Πολιτών ζήτησε την ε, νέα καταμέτρηση των ψήφων στα Τύρανα ώστε να ληφθούν υπόψη οι λανθασμένες ψήφοι, δηλαδή οι ψήφοι ε, που τοποθετήθηκαν σε, σε λάθος κάλπες για την εκλογή των δημάρχων. Ε, Η απόφαση αυτή τελικά ελήφθη, αλλά υπήρξαν και αντιρρήσεις, γιατί η καθυστέρηση ανακοίνωσης ε, του εκλογικού αποτελέσματος για τα τύρανα συνεχίστηκε και η κατάσταση ε, γινόταν όλο και πιο τεταμένη, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση της ΟΑΣΕ για νέα καταμέτρηση των ψήφων στα Τύρανα, η αντιπολίτευση απειλεί να αποσυρθεί από το Κοινοβούλιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέσβη Σέκη και πρέσβη ε, Όρβης από τη ΣΥΠΑ άρχισαν ε, και ξεκολουθούν να κάνουν ε, την διπλωματία του έλα μιλώντας και συναντώντας τους ηγέτες το όλων των πολιτικών κομμάτων ζητώντας να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Η ΟΑΣΕΑ από τη Δευτέρα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα και για τα τύρανα όπου ο Ρούζικ Μπάσα κέρδισε με διαφορά 81 ψήφων. Από τη Δευτέρα και μετά όλα τα κόμματα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονα. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το εκλογικό σώμα των εποπτών ε, των τυράννων και αυτή η απόφαση θα είναι και τελεσίδικη. Η εκλογική διαδικασία δηλαδή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Κύριε Πρόεδρε, κάποιες παρατηρήσεις που εκφράζουν τώρα την προσωπική μου γνώμη. Όλοι γνωρίζουμε πως η κατάσταση στην Αλβανία εδώ και χρόνια ε, χαρακτηρίζεται από βαθιά πολιτική δυσπιστία και μεγάλη πόληση, πόλωση των, της πολιτικής και της κοινωνίας. Η συμμετοχή των Αλβανών στις εκλογές δείχνει πως ο κόσμος ενδιαφέρεται για τη χώρα του και για το μέλλον του, της. Αυτές λοιπόν οι εκλογές θα έπρεπε να έχουν δείξει πολιτική οριμότητα των Αλβανών ηγετών και την ικανότητά τους να διεξάγουν εκλογές σύμμορφες με ψηλές διεθνείς προδιαγραφές. Δυστυχώς όμως εντύπωση μου είναι ότι η επιδείνωση της εκλογικής κατάστασης έδειξε και πάλι τα μόνιμα προβλήματα της αλβανικής πολιτικής και της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας. Είναι, πρόκειται για την ανικανότητα να διεξάγει πολιτικό διάλογο, να εξεύρει συναντικές λύσεις και να συμφωνήσει για βασικές δημοκρατικές αρχές. Εγώ φοβούμαι και ανησυχώ ότι οι εκλογές δεν θα βοηθήσουν την Αλβανία να ξεπεράσει το πολιτικό τέλμα. Ξέρω πως ακούγομαι απεσιόδοξο. Φυσικά το χειρότερο σενάριο θα είναι αν παραταθεί το πολιτικό τέλμα. Γνωρίζω πως ακούγομαι απεσιόδοξο, αλλά θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής αν οι μελλοντικές εξελίξεις με αποδείξουν λάθος, να ότι έχω κάνω λάθος, γιατί εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον αλβανικό λαό. Το νομικό τμήμα τώρα ε, του εκλογικού νόμου θα ε, προκαλεί κάποιες απορίες, αλλά αυτό θα πρέπει να αφαιθεί στους εμπειρογνώμονες και στα κατάλληλα θεσμικά όργανα. Η πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια της χώρας εξαρτάται από τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς ηγέτες. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν σε αυτή, τι αυτές τις συνθήκες το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει μόνο αν μιλάμε μια φωνή και αν αυτή η φωνή είναι συντονισμένη με αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα της χώρας και του λαού της, γιατί είμαι πεπισμένος πως οι Αλβανοί αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο σκιώδεις συζητητές. Μιχαήλ Τρεμόπουλος και ο κύριος Χουντής είναι στον κατάλογό μου. Ο Μιχαήλ Τρεμόπουλος. Μα δεν είναι. Και ο κύριος Κασουλίδης μετά. Το λόγο έχει ο κύριος Τρεμόπουλος. Και μετά ο κύριος Χουντής. Ε, ήμουν ε, ένας από αυτούς που βρίσκονταν εκεί ως παρατηρητές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εκλογές της ε, Αλβανίας, στις τοπικές εκλογές. Είχα τη δυνατότητα να κάνω μια σύγκριση με παλιότερες εποχές, μια και πήγα μετά το 90 αρκετές φορές και σε εκλογές του 1993. Ε, πραγματικά αυτό που έχω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Κουκάν, ε, είναι κάποια επιμέρους στοιχεία, μια και μαζί πηγαίναμε ε, στα οικολογικά τμήματα, μέσα στα τύρανα και έξω από αυτά. Το βασικό μου συμπέρασμα είναι ότι στην Αλβανία χρειάζονται να γίνουν αρκετά βήματα ακόμη για να ξεπεράσουν ε, του παρελθόντος την ε, κυριαρχία της οικογένειας ή της φάρας και να μετριαστούν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να περάσουν δηλαδή σε μια πραγματική πολιτική κοινωνία και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Μερικά σημεία τα οποία έχω να προσθέσω από την εμπειρία και τα οποία είδαμε μαζί με τον κύριο Κουγκάν και, τους, και τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Είδαμε να υπάρχουν αφήσει οι οποίες καλούσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την οικογενειακή ψήφο. Αυτό φαίνεται περίεργο για κάποιον πολίτη άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη, αυτό που είδαμε είναι μία περίπτωση και μας εξήγησαν ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ περισσότερες φορές ο πατέρας, ο αρχηγός της οικογένειας να πηγαίνει με τρεις ταυτότητες για να ψηφίσει για όλη την οικογένεια. Τα τμήματα, τα εκλογικά ήταν μεικτά. Ε, αυτό ο, σήμαινε ότι ήταν κάποια αναλόγια όπου φαινόταν οι, ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι την ώρα που ψήφισαν ήταν πολύ κοντά και μπορούσε να ψηφίζει ταυτόχρονα ο σύζυγος με τη σύζυγο, να συνεννοούνται τι θα ψηφίσει και πού θα βάλει σταυρό ή να είναι ο, γιο, ε, γιος ή η κόρη. Ο επηρεασμό δηλαδή ακόμη και την τελευταία στιγμή. Είδαμε επίσης και ενημερωθήκαμε για τις απαγορεύσεις χρήσης κινητών τηλεφώνων την ώρα της ε, ψηφοφορίας. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ψηφοφόρου να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο είτε για να συνομιλούν εκείνη τη στιγμή, είτε για να φωτογραφίζουν το ψηφοδέλτιο, το οποίο στη συνέχεια είχαν τη δυνατότητα να επιδείξουν, επειδή ένα είναι το ψηφοδέλτιο, ήταν η συγκεντρωτική η παρουσίαση των κομμάτων, με το σταυρό στο κόμμα στο, για το οποίο έχουν συνοηθεί να ψηφίσουν και τη φωτογραφία αυτή να την επιδείξουν μετά στον κομματάρχη, στον προϊστάμενο μιας υπηρεσίας ή και στον ιδιώτη εργοδότη. Επίσης ε, ενημερωθήκαμε ότι και υπήρχε ένα σημάδι με μελάνι στο δάχτυλο ε, το οποίο μας είπαν ότι είναι ανεξίτηλο και εμπόδιζε το να ξαναψηφίσουν οι ίδιοι άνθρωποι σε άλλο εκλογικό τμήμα. Στο πρώτο τμήμα που μπήκαμε, βλέπαμε να φεύγουν χωρίς το σημάδι. Ρωτήσαμε τι συμβαίνει, μας απάντησε κάποιος ότι η μελάνη είναι αόρατη. Ε, αποδείχθηκε ότι απλώς είχαν ξεχάσει. Στο επόμενο τμήμα που μπήκαμε, προσωπικά είχα την ευκαιρία, ζήτησα, να μου βάλουν και μένα ένα σημάδι. Μου το έβαλαν. Μέσα σε δέκα λεπτά, με απλή χρήση του σάλιου, το είχα βγάλει. Και θεωρητικά θα μπορούσα, αν ήθελα να καταστρατηγήσω τη διαδικασία, να πάω κάπου αλλού. Άλλοι, όπως ο κύριος Κουκάν που το έβαλε, αλλά δεν το προσπάθησε αμέσως, έμεινε και την υπόλοιπη μέρα. Σας δίνω λοιπόν μερικές ε, φωτογραφίες ε, μιας εμπειρίας που είχαμε εκεί στην, ε, στην περιοχή για να καταλάβετε και τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Ο καθένας μπορεί να αμφισβητήσει το, το αποτέλεσμα και η αντίδρασή του αυτή να βρει ευρύτερα οπαδούς υπάρχει μια πολύπλοκη διαδικασία που δεν την έχω συναντήσει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετεί υποτίθεται την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων αλλά τελικά δεν νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι στην ίδια την πολιτική κουλτούρα και γι' αυτό ελπίζω ότι θα γίνουν βήματα μέσα στο επόμενο διάστημα ούτως ώστε να μπορέσει ε, αυτή η χώρα να έχει μια πραγματική ευρωπαϊκή προοπτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Το 1993 ήμουν και εγώ. Μάλλον και οι δυο μας θα ήμασταν πολύ πιο νέοι. <laughs> Αλλά ήμασταν εκεί στις εκλογές στην Αλβανία. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Χουντής της Γκουε, που είναι εισηγητής για την Αλβανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν, τον κύριο Τρεμόπουλο και όλους τους συναδέλφους που ως αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρακολούθησαν τις πρόσφατες εκλογές στην Αλβανία ως παρατηρητές. Μας έδωσαν κάποιες εικόνες. Από εκεί βγαίνουν δύο συμπεράσματα κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο, καλό είναι αυτό το σύστημα. Συζητούσαμε και χτες το θέμα των εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες προκειμένου να διαπιστώσουν την αντικειμενικότητα αυτής της διαδικασίας αλλά όπως διαπιστώσαμε αυτό το σύστημα έχει τα όρια του. Ο κύριος Κούκαν, ο κύριος Τρεμόπουλος και οι τρεις ακόμα συνάδελφοι δεν μπορούσαν <laughs> να λύσουν ή να έχουν συνολική εικόνα αυτού του προβλήματος καλή παρουσία τους, έδινε ένα κύρος, αλλά έχει και κάποια όρια αυτή η διαδικασία. Και το δεύτερο, οι εικόνες που μας αναφέρθηκαν για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας είναι η μια πτυχή του προβλήματος. Από ό,τι είδαμε μετά, το κακό παραμονεύει και σε άλλες φάσεις της εκλογικής διαδικασίας μέχρι που να εκδοθούν αδιάβλητα, αντικειμενικά και κοινώ παραδεκτά αποτελέσματα. Επομένως θα έλεγα η συμβουλή, βεβαίως είναι θέμα της, των αλβανικών πολιτικών δυνάμων, μιας απλοποίησης της εκλογικής νομοθεσίας, διότι αν αυτό συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε εκλογές στην Αλβανία, καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγει ποτέ από την πολιτική ένταση, ιδιαίτερα όταν αμφισβητούνται τα εκλογικά αποτελέσματα όπου μιλάει ο λαός. Και το τρίτο, είναι ότι πραγματικά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στον τομέα του εκδημοκρατισμού, της πολιτικής ζωής των, ε, στην, ε, γειτονική, ε, στην Αλβανία, προκειμένου να πούμε ότι έχει προετοιμαστεί καλά ή, εν πάση περιπτώσει, σε όφελος του λαού προσβλέπει στην ένταξη στην ευρωπαϊκή προπτυγή. Το δεύτερο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, είναι να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να αφήσουν ανοιχτή την πρόσκληση και την προπτική της ευρωπαϊκής προπτικής της Αλβανίας επισημένοντας ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Πρέπει να γίνουν σοβαρά πράγματα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς κουραστικά αποδίδοντας ευθύνες σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και κυρίως στις δύο μεγαλύτερες, να προσπαθήσουν να υπάρξει μια συνονόηση, ένας σεβασμός, ένας πολιτικός διάλογος για να βγει η χώρα από τα διέξοδο. Επισημαίνω ότι δυστυχώς οι δημοτικές εκλογές δεν άμβληναν την πολιτική κρίση, αντίθετα όπως είπε και ο κύριος Κούκαν, μάλλον την ενέτειναν και προσθέτω αγαπητοί συνάδελφοι ότι στον ορίζοντα έρχονται σημάδια και οικονομικής κρίσης και οικονομικής κρίσης στην Αλβανία, λόγω και προβλημάτων εσωτερικά οικονομικών, αλλά λόγω του ότι πληρώνει και θα πληρώσει τις συνέπειες της κρίσης γειτονικών χωρών, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, πράγμα που σημαίνει πολιτική κρίση και οικονομική κρίση, το μείγμα θα είναι εκρηκτικό. Επομένως, η εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης να αμβληθούν αυτές οι εντάσεις το γρηγορότερο δυνατό, ως έκκληση και με κάθε τρόπο βοήθεια, βοήθεια επαναλαμβάνω από τη δική μας την πλευρά, είναι η καλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στον αλβανικό λαό. Ευχαριστώ. Grazie, la parola al collega Σας ευχαριστώ, ο συνάδελφος Μποστινάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους σας για την υποστήριξη, για την αλληλεγγύη που μου δείξατε όταν δέχθηκα επίθεση από έναν Αλβανό ομιλητή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα το προνόμιο να λάβω επιστολή από τον ίδιο τον πρόεδρο Μπούζεκ προσωπικά, ο οποίος καταγγέλει και καταδικάζει στην απαράπτη, συμπεριφορά της κυρίας το πάλι συγκεκριμένα της Προέδρου του Κοινοβουλίου. Που, και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπούζεκ για τον τρόπο που φέρθηκε και την ποιότητα της δήλωσής του. Τώρα ερχόμενοι στα γεγονότα και στις εξελίξεις στην Αλβανία. Ενδιάμεση έκθεση, ε, προσωρινή έκθεση του ΑΣΕ. Μία πρόταση θα σας αναφέρω ε, στις 8 ε, Μαΐου. Παρότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, άρχισαν να ανοίγουν οι κάλπες που είχαν εντοπιστεί στο αίτημα και να καταμετρά τις ε, ψήφους, τα ψηφοδέλτια για το Δήμο των Τύραμ. Νομική βάση για να ανοίξουν οι κάλπες δεν ήταν σαφής. Unclear λέει στα αγγλικά. ήταν ασαφής λοιπόν οι λόγοι για τον ΟΑΣΕ. Χθε έγινε μια γνωστή δήλωση ε, γνωστή δήλωση από την κυρία Άστον και τον Επίτροπο Φιούλε που επανέλαβαν ουσιαστικά την πρόταση με άλλα λόγια νομική ευρωστία της απόφασης ε, για να μετρήσει αυτές τις χαμένες κατά κάποιο τρόπο κάλπες είναι ένας λόγος ανησυχίας. και θεωρεί ότι η διαδικασία προσφυγής θα πρέπει να είναι διαφανής, δίκαιη και να διεξαχθεί ανεξάρτητα και σε πλήρη συμμόρφωση με το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Σας καλώ όλους τώρα Όταν είχαμε μιλήσει για, είχαμε ζητήσει να ανοίξουν οι κάλπες, μας είχε πει ο κύριος Μπερίσα ότι είναι, αντι, ε, είναι απαράδεκτο και ότι το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο το προβλέπει. Ζήτω το Σύνταγμα είχαμε πει, το δεχθήκαμε. Το Σύνταγμα είναι το θεμελιώδη νομοθέτημα κάθε δημοκρατικής χώρας. Τώρα όμως δεν ισχύει αυτό. Η κυβέρνηση αποφάσισε να ξανανοίξει τα, τις κάλπες, όχι όλων των εκλογικών τμήματων των τυράων, αλλά κάποιες, από κάποια εκλογικά τμήματα που είχαμε κάποιους ισχυρισμού για να ίσως ε, επικρατήσει ένα συγκεκριμένο κόμμα. Και θα ήθελα εδώ να σας παρακαλήσω να λάβετε υπόψη σας το ότι δεν έχουν προηγούμενο αυτές οι όλες οι διαδικασίες. Για ποιο λόγο, γιατί σε ένα εκλογικό τμήμα βρήκαν πάνω από 200 200 ψηφοδέλτια, περισσότερα από τους ψηφοφόρους που ήταν εγγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Θαύμα πρέπει να έγινε εκεί λοιπόν. Δηλαδή τι κάναν, βάλαν στην ίδια κάλπη ε, ψηφοδέλτια που ήταν για το Δήμαρχο, για το Δημοτικό Συμβούλιο των Τυράννων ή για τα μικρά συμβούλια, για τα, τα τις λεγόμενες επαρχίες, μικρότερες διοικητικές περιφέρειες. Όλα αυτά στο ίδιο καλάθι εντός αγωγικών χωρίς κανένα, καμία νομική αιτιολόγηση. Και τέλος σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας και να λάβετε υπόψη σας και τα σοφά λόγια του κυρίου Κούκαν. Τι μπορούμε να κάνουμε πλέον για να αποφύγουμε μία μείζωνα κρίση. Είπε ένα πολιτικό Αλβανίας ότι μπορεί να υπάρξει εμφύλιο στην Αλβανία και σας παραπέμπω στα λόγια αυτά. Λοιπόν, πρέπει η Ευρώπη να μιλήσει με μία φωνή, μαζί με την Κομισιόν και να ζητήσουμε οποιαδήποτε απόφαση να σέβεται και να τηρεί πλήρως όλες τις ε, υφιστάμενες νομικές διατάξεις και τίποτε άλλο. Μόνο τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις, και συνταγματικές διατάξεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουμε ανεφόρο να στηρίζουμε τη μία πλευρά και ίσως έτσι ενθαρρύνουμε την άλλη πλευρά να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να προχωρήσει σε κλιμάκωση της κατάστασης. Άρα να έχουμε ε, βιοπραγίες και να μην μπω και φίλιο πόλεμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την αλληλεγγύη που μου δείξατε πολλοί από εσάς απέναντι στην επίθεση της Προέδρου του Αλβανικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Kasoulidis. You have the floor. Ο κύριος Κασουλίδης τώρα το λόγο. Yes, thank you, Chairman. It is obvious that um, στην Αλβανία υπάρχει πολύ έντονη πόλωση. Και επίσης τα δύο μεγαλύτερα κόμματα είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Κάθε ψήφος μετράει λοιπόν. Αντί να μιλάμε για τις ευθύνες των δύο πλευρών, αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει κάποια ευθύνη των υπηρεσιών που συμβουλεύουν για τη διεξαγωγή των εκλογών. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αναρωτιέμαι πώς γίνεται και δεν τους συμβούλεψαν για το χρώμα του ψηφοδελτίου που θα έπρεπε να είναι διαφορετικό για τις δημοτικές και διαφορετικό για, ε, ε, για το Δήμαρχο και διαφορετικό για το Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς γίνεται δηλαδή ο πρόεδρος να επιτρέψει ε, ένας εκλογέας να ρίξει στην κάλπη δύο ψηφοδέλτια, είτε ήταν για το Δήμαρχο ή για το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, σε εκείνο το σημείο και μόνο θα μπορούσε να αποφευθεί το λάθος. Τρίτον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο μας, δεν νομίζω ότι εξυπηρετούμε καλή υπόθεση αν επιτρέψουμε να γίνουμε εμείς κριτές ε, που θα ευνοήσουν τη μία ή την άλλη πλευρά. Αν το κάνουμε αυτό θα ρίξουμε λάδι στη φωτιά και δεν θα βοηθήσουμε τον λαό της Αλβανίας ούτε το μέλλον της χώρας. Τα επιχειρήματα γιατί τώρα έτσι και γιατί την άλλη φορά αλλιώς ε, όταν άνοιξαν οι κάλπες κλπ. Ας τα αφήσουμε αυτά να τα κρίνουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές και ελπίζω ότι το δικαστικό σύστημα τουλάχιστον λειτουργεί στην Αλβανία. Αλλιώς τι νόημα έχει να μιλάμε για υποψηφιότητα στην, ε, και προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ευχαριστώ. Μετά τα σχόλια που άκουσα πολύ προσεκτικά, επαναλαμβάνω τη θέση της ομάδας μας, ε, την αντιπολίτευση, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρχήν δεν πρέπει να παρακολουθεί τοπικές εκλογές. Ε, έχω κάθε σεβασμό στον ε, πρόεδρο Κούκαν και τον Προεδρείο, αλλά ήταν λάθος ενδογενές στην απόφαση τι νόημα έχει η αντιπροσωπεία. Οι τοπικές εκλογές πρέπει να παρακολουθούνται από την Επιτροπή Περιφερειών ή το Συμβούλιο της Ευρώπης και εμείς πρέπει μόνο βουλευτικές εκλογές και προεδρικές. Εμείς δεν είμαστε τοπικοί ε, παράγοντες και άρχοντες, είμαστε ε, εθνικοί παντού γίνονται. Εμείς δεν είμαστε μέλη τοπικών δημοτικών συμβουλίων. Ε, τώρα, πώς ε, νομιμοποιούμε τα αποτελέσματα, πώς ενθαρρύνουμε τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, πώς προάγουμε την συμφιλίωση μεταξύ των πολλωμένων ε, κομμάτων. Δεν τα καταφέραμε, αρνητικό είναι το, αποτέλεσμα. Ε, δηλαδή, τώρα είδαμε διαφορετικά την Αλβανία ως υποψήφια. Όχι. Εγώ θα πάω στη στη για να πάω να συμμετάσχω σε Μακεδονία υπομιλήτης ε, για να, δω, να δούμε πώς ε, δεν ε, πήγαν παρατηρητές στη γειτονική χώρα Μακεδονία λέει ο μιλητής γιατί δηλαδή πήγαμε να παρακολουθήσουμε τοπικέ εκλογές στην Αλβανία και δεν πήγαμε να βοηθήσουμε την ευάλωτη χώρα Μακεδονία κατά τον ομιλητή. Ο κύριος Κουμουτσάκος. ήμουνα και εγώ μέλος της Επιτροπής ε, της που επισκέφθηκε την Αλβανία από την οποία φύγαμε στις 9 Μαΐου. Η μέρα που είχαν ήδη κλείσει κάλπες ήταν μία μέρα μετά. Σήμερα, 15 ολόκληρες μέρες μετά, έχουμε μία ιδέα για το αποτέλεσμα που φαίνεται ότι είναι η οριστική. Μεσολάβησαν 15 ημέρες καταμέτρησης. Και αυτό από μόνο του κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάλφοι είναι ενδεικτικό του πόσο όριμη είναι η εκλογική διαδικασία στην Αλβανία. Και δεν χρειάζεται κανείς να επεκταθεί σε ειδικέ λεπτομέρειες όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Κασουλίδης. Ανεξάρτητα λοιπόν από το πώς αξιολογούμε τις επιμέρους πτυχές της εκλογικής διαδικασίας, δεν μπορεί παρά να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό συμπέρασμα. Η Αλβανία δεν είναι πλέον μια νεοπαγής δημοκρατία. Μετράει σχεδόν μία δεκαετία και. Και αυτό το στοιχείο του χρόνου δεν μπορούμε να τα αγνοούμε στις αξιολογήσεις μας. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ποιότητα της λειτουργίας βασικών πτυχών της δημοκρατικής διαδικασίας και του πολιτεύματος δεν λειτουργούν επαρκώς και πάντως δεν λειτουργούν ικανοποιητικά με τις δικές μας αξιολογήσεις και με τα δικά μας standards. Και αυτό δεν μπορούμε παρά να το υπογραμμίσουμε. Γιατί θα δούμε και πρέπει να δούμε και να παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση από εδώ και πέρα στη χώρα αυτή. Οι εντάσεις και η πόλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όσον αφορά αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τάνο, κατά πόσο έπρεπε να είμαστε παρόντες ή όχι, είναι βέβαιον και όλα όσα είπα και όλα όσα συζητήθηκαν πριν, ότι έπρεπε να είμαστε παρόντες για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Αλβανία, η οποία διεκδικεί να ξεκινήσει ενταξιακή διαδικασία στην Ένωση. Κλείνω με ένα μόνο σημείο, κύριε Πρόεδρε. Η αποστολή των παρατηρητών πολύ σωστά αποφάσισε να στείλει παρατηρητές και στην Χιμάρα. Μια περιοχή όπου στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί εντάσεις τέτοιες που είχαν οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο ανθρώπων. Είναι ελπιδοφόρο ότι στις εκλογές αυτές δεν παρατηρήθηκαν τέτοιες εντάσεις και δεν υπήρξαν παράπονα ή ενστάσεις για τον τρόπο που διεξήχθηκε η ψηφοφορία. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς στην Αλβανία γιατί θα πρέπει οι ψήφοι τους που δίδονται σε τοπικό επίπεδο να μεταφέρονται με κάλπες σε κάποιο κεντρικό σημείο καταμέτρησης, μακριά από τον τόπο εκλογής. Η απάντηση των αλβανικών αρχών σε αυτό είναι ότι προτιμούμε να την ελέγχουμε κεντρικά τη διαδικασία, διότι στα επιμέρους εκλογικά τμήματα είναι πιο δύσκολο να ελέγξουμε αν υπάρχουν παρατυπίες, παρανομίες, αλλίωση ψηφοφορίας. Αυτή και μόνο η παραδοχή είναι ένα πρόσθετο σημείο προβληματισμού και έντονης ανησυχίας εκ μέρου μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούκαν για να, πει τον τελευταίο, να έχει τον τελευταίο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρεις φράσεις μόνο. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη σύντομη συζήτηση. Εκτιμώ ε, όλος ιδιαίτερο τα περαιτέρω στοιχεία που έδωσαν ως ενημέρωση οι συνάδελφοι που ήταν μαζί μου στην αποστολή. Συμφωνώ με τον κύριο Κασουλίου ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ούτε κριτές, ε, ούτε τιμητές, ε, ούτε να αξιολογούμε τις εκλογικές διαδικασίες στην Αλβανία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επαναλαμβάνω βέβαια αυτό που είπα Και είναι ένα άλλο θέμα που θέλω πάλι να στηρίξω και να συμφωνήσω με τον κύριο Κασουλίδη. Δεν πρέπει να μπούμε σε ε, κάποια αντιπαράθεση δεν θα ήταν καλό και θα εμβάθυνα ακόμη περισσότερο τις εντάσεις. Πρέπει να μιλήσουμε πράγματι με μία φωνή, ε, να είμαστε ε, νιαίοι στη στάση μας και στο λόγο μας. Φυσικά και δεν υπάρχει αφιβολία ότι η κυβέρνηση το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε καλή δουλειά για την προετοιμασία των εκλογών. Και όπως σας είπα, δεν είμαστε δυσαρεστημένοι για το πώς πήγε η ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα που άρχισε η διαδικασία καταμέτρησης και είναι και η αποδοχή των αποτελεσμάτων των εκλογών. Εκεί είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι και φοβάμαι ότι θα δούμε την ίδια κατάσταση μετά τις κοινοβουλευτικές, τις βουλευτικές εκλογές του Ιωνίου του 9. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Μια χώρα που στην τελευταία έκθεση προόδου ε, δεν πήρε καν το καθεστώς χώρας υποψήφιας ε, και αν αυτή η εσωτερική κρίση ε, παραταθεί, επιμηκυνθεί, αυτό θα είναι κακό για τη χώρα και θα είναι κακό και για το λαό βέβαια της Αλβανίας όπως προείπα. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί πρωτίστως. Σε ό,τι αφορά τώρα τις παρατηρήσεις του Charles Τάνοκ. Πριν ληφθεί η απόφαση για την αποστολή αντιπροσωπεία στην Αλβανία, συζητήθηκε και δεν υπήρξε ομοφωνία. Ελήφθη πάντως η απόφαση και το ίδιο ακριβώς ίσχυε και για την μία αποστολή αντιπροσωπείας εκλογές στη Μακεδονία, λέει ο ε, υπήρχε πάντως ανάγκη να γίνει συζήτηση, βαθιά συζήτηση, σε βάθος συζήτηση. Αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής ήταν να μείνουμε στους ισχύοντες κανόνες ή ετέθηκε το ερώτημα αν θα έπρεπε να, κάποιες φορές να, να υπάρχουν εξαιρέσει για τις αποστολές ε, αντιπροσωπιών παρατήρησης εκλογών. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο αφορά την ώρα των ερωτήσεων για την ΕΕΔ, Ο συνάδελφος Καμίνσκι όμως δεν είναι εδώ, γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε, οπότε διακόπτουμε για 10 λεπτά.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 Bene, Ώρα των ερωτήσεων. Προς την ε, ΕΙΕΔ που θα αφιερωθεί και αφορά τον εκδότη Άντριου Βέτσμπουρτς στη Λευκορωσία. Εφόσον η απάντηση του ΣΥΠΑ της εκπροσώπου δεν ήρθε στη, μέσα στι έξι εβδομάδε που προβλέπονται. Ο κύριο Καμίνσκι ζήτησε να συμπεριληφθεί αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη τη συναντησή μα. Οπότε ο κύριο Καμίνσκι έχει το λόγο για να παρουσιάσει τα ερωτήματά του και να πάρει και τι απαντήσει του από πλευρά τη εξωτερική υπηρεσία δράση από τον κύριο Μάικη. Κύριε Καμίνσκι, έχετε το λόγο. Microphone. E, e, κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει 50 ημέρε από τη φυλάξη του κύριου Πότομπουκ. Στι 11 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα καταδικάστηκε σε 15 ημέρε φυλάκιση από το δικαστήριο τη Λευκορωσία με Υποτιθέμενη την κατηγορία της συμμετείχε στις 19 ε, Δεκεμβρίου σε μια διαδήλωση στο Μίνσκ. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι είχε ενεργό συμμετοχή στη διαδήλωση αυτή, παρότι ο ίδιος λέει ότι απλά ασκούσε τα δημοσιογραφικά του καθήκοντα και την εκδοσή, εκδοχή του ε, την επιβεβαίωση επιβεβαίωσε η πολωνική κοινότητα, μέλος ενεργό της οποίας είναι στην Λευκορωσία. οι λευκορωσικές αρχές ε, προσπάθησαν να επιμηκύνουν, να παρατείνουν την κράτησή τους στις φυλακές. Και αυτό επιβεβαιώνεται, εφόσον πλέον είναι 50 μέρες στη φυλακή ήδη. Εξού και το ερώτημα που θέτω στην Επιτροπή. Είπατε εκπρόσωπος. Έχει γνώση. Και τι δράση θα αναλάβουν. Αυτά έλεγε και η ερώτησή μου τόσο Άλλος, Μάλιστα, την απάντηση θα μας δώσει ο κ. Ματής από την ε, ΕΙΕΔ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, θα ήθελα να σα πω ότι εξ όσων γνωρίζουμε είναι η πρώτη φορά που υπάρχει γύρω σε ερωτήσεων προ την ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση στην Επιτροπή ΑΦΕΤ εδώ και χρόνια ε, δεν είχαμε λάβει ερωτήσεις από την Επιτροπή σας. Δεν έχουμε ακόμη συμφωνήσει τους όρους, ε, πώς δηλαδή θα διεξάγεται η διαδικασία αυτή των ερωτήσεων στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης από την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε εκπονήσει τους σχετικούς κανονισμούς. Πάντως η Εξωτερική Υπηρεσία είναι έτοιμη να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα του εξώτημου βουλευτού κ. Καμίνσκι. Πρέπει Ωστόσο, να σας μιλήσω λίγο για τη διαδικασία. Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλαξε τον εσωτερικό του κανονισμό, ούτω ώστε οι βουλευτές να μπορούν να απευθύνουν ερωτήσει απευθεία ε, στην υπάτη εκπρόσωπο για την ε, ΚΕΠΑ. Πρόκειται για το νέο κανόνα 117 παράγραφος 1. Μία πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τι νέε θεσμικέ διευθετήσεις υπό τη συνθήκη τη Λισαβόνη. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο συνεχίζονται οι γραπτές νοβλευτικές ερωτήσεις να απευθύνονται μόνο στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Εδώ μιλώ εξ ονόματος ε, της ΕΙΕΔ, αλλά ο κύριος Καμίνσκι υπέβαλε την ερώτησή του την 1η Μαρτίου στο Συμβούλιο. Άρα εμείς έπρεπε ως υπηρετησία εξωτερικής δράσης να στραφούμε στο Συμβούλιο για να μάθουμε τι συμβαίνει. Η απάντηση που λάβαμε από το Συμβούλιο, στο οποίο απευθυνόταν η ερώτηση, ήταν ότι όλες οι ερωτήσεις, μάλλον, συγγνώμη, όλες οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που απευθύνονται επισήμως στο Συμβούλιο, ακόμη και αν είναι καθαρά διαδικαστικής φύσεως, πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Σε επίπεδο υπουργών δηλαδή. Σε αντίθεση με τι ερωτήσει που απευθύνονται στην Κομισιόν, δεν μπορούν να μεταβιβάζονται απλά στην υπατή ούτε μπορεί να μπορεί το Συμβούλιο να απαντά στη θέση της ΥΠΑΤΣ εκπροσώπου, τις οποίες τα καθήκοντα υπερβαίνουν αυτά του Υπουργείου Εξωτερικών Θεμάτων. Αυτά μας είπε το Συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και αυτό εξηγεί το λόγο για τον οποίο δεν λάβατε νωρίτερα απάντηση στην ερώτησή σας. Η αντιμετώπιση, μάλλον η υποβολή των ερωτήσεών σας άμεσα στο μέλλον, στην απευθεία στην υπηρεσία μας, ε, θα έχει και ως αποτέλεσμα την ταχύτερη απάντησή τους. Το Συμβούλιο απάντησε πάντως ε, στις 28 Απριλίου του τρέχοντος στον ε, κύριο Καμνισκή και λέει στην απάντησή του. Επειδή πρόκειται για ερώτημα προς την υπατή εκπρόσωπο για την ΚΕΠΑ. το Συμβούλιο παρακαλεί τον εξώτομο βουλευτή να υποβάλει το ερώτημά του απευθεία στην υπατή εκπρόσωπο όπω προβλέπετε στο άρθρο 117 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Ήρθαμε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε κατά πόσον ε, είναι δυνατόν οι βουλευτές να απευθύνονται ε, απευθείας στην κυρία Άστον και να της υποβάλουν ερωτήσεις. Χθε το βράδυ επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι ακόμη δεν είναι δυνατόν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου να ε, ρωτούν απευθείας την κυρία Άστον. Πάντως γίνονται κάποιες εργασίες και έχω και ένα υπόδειγμα του δελτίου που θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε στο μέλλον όταν θέλετε και θα μπορείτε πλέον να υποβάλλετε ερωτήσεις όχι μόνο πια στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή αλλά και στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και αντιπρόσωπο της Επιτροπής αλλά και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ενημέρωση που λάβαμε όμως είναι ότι δεν είναι ακόμη επιχειρησιακό, δεν λειτουργεί ακόμη αυτό το σύστημα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν λειτουργεί ακόμη αυτό το σύστημα δεν είναι δυνατόν να υποβάλλετε απευθεία ερωτήσεις στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο. Είναι θέμα εβδομάδων πάντως από ό,τι καταλαβαίνω. Και ελπίζω να μπορέσουμε να αποφύγουμε καταστάσεις σαν τη Να πω, επειδή θέλω να ε, δώσω και λίγη ουσία στην απάντησή μου και συγγνώμη που δαπάνησα τόσο χρόνο για να σας μιλήσω για τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό και καταλαβαίνει, πρέπει να καταλάβει και ο κ. και, και οι υπόλοιποι τι συμβαίνει. Όταν λοιπόν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, Μελετήσαμε την ερώτηση και είπατε εκπρόσωπο τώρα έχει απαντήσει την ερώτηση του κ. Καμίνσκι. Η οποία συνοδεύτηκε ε, από μια επιστολή την οποία υπογράφει ο αναπληρωτή Γενικός Γραμματέας κ. Ποπόφσκι και εστάλει χθε στον κύριο Καμίνσκι. Μίλησα με τον ε, κύριο Καμίνσκι που μου λέει ότι δεν το έχει λάβει ακόμη το γράμμα αυτό που ε, εστάλει χθε στο γραφείο του. Μπορώ να του το δώσω, να του το εγχειρήσω αυτή τη στιγμή. Ευχαρίστω, αλλά μπορώ και να διαβάσω την ε, απάντηση στο αρχικό ερώτημα τη 1 η Μαρτίου. Αλλά είναι και ενημερωμένοι, επικαιροποιημένοι με στοιχεία ε, τα οποία έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Αν σας ενδιαφέρει κύριε Καμίσκη, είτε μπορώ να σας το διαβάσω ε, τώρα μεγαλοφόνος, είτε να δώσω την επιστολή στον κύριο Καμίνσκι προσωπικά. Κύριε Καμίνσκι, τι επιθυμείτε, πώς επιθυμείτε να λάβετε την απάντηση. Πρόεδρε, πιστεύω πως το θέμα που συζητάμε σήμερα, τη Λευκορωσία δηλαδή, όχι τα διαδικαστικά θέματα, είναι τόσο σημαντικό που πιστεύω πως θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε ώστε να γραφεί στα πρακτικά τα όσα έχει να μας πει ο αξιότιμος εκπρόσωπος της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το θέμα αυτό του κ. Ποτσόπος που εξακολουθεί να είναι υποκράτηση και για την ίδια τη Λευκορωσία. Οπότε ευχαρίστως να ακούσω τον ε, φίλο μας από την Εξωτερική Υπηρεσία αν μπορεί να διαβάσει την επιστολή. Αυτό επιθυμεί ο κ. Καμίνσκι λοιπόν. Ναι, εγώ είμαι ο κ. Καμίνσκι και μόλις εξέφρασα τη θέλησή μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά και θα κάνουμε αυτό που μας ζητά ο αξιότιμος κύριος Βουλευτής. Θα σας διαβάσω τώρα την απάντηση της Αντιπροέδρου, είπα της εκπροσώπου κάθε άστον, όπως διαβιβάστηκε στον κύριο Καμίσκι. Η είπα τους εκπρόσωπους ευχαριστεί τον κύριο Βουλευτή γιατί τονίζει την πίεση που δέχονται οι... Ε, αντιπολιτευόμενοι και εκπρόσωποι της ε, κοινωνίας των πολιτών στην Λευκορωσία και ε, ευχαρίστω μπορεί να σας ενημερώσει για την κατάσταση του κύριου Πογόβους, ε, για τον, τον ανταποκριτή της πολωνικής εφημερίδας και έχει ως εξή. την 1η Ιανουαρία, Ιανουαρίου οι πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας της Λευκορωσίας και ζητώ συγγνώμη αν δεν ε, λέω σωστά το όνομα ε, των Πόλων, ε, έφεραν στο δικαστήριο το Μίνσκ τον κύριο Πόκοσαν πλήρωσαν 250 ευρώ εκεί οι αντιπολιτευόμενοι και απελευθερώθηκε η εισαγγελία του Μίσκ θεώρησε ότι η ποινή αυτή ήταν πολύ ήπια. Στη συνέχεια το ανώτερο δικαστήριο του ΜΙΣΚ καταδίκασε τον κύριο Πόκουβς σε 15 μέρες φυλάκισης για συμμετοχή σε διαδηλώσεις που ήταν απαγορευμένος μετά από τις προεδρικές εκλογές. Ο κύριο Ποσκόμποτς κάλυπτε τις διαμαρτυρίες αυτές για την καζέτα Βιμπόσκα, την πολωνική καθημερινή εφημερίδα. Σύμφωνα με την, τις πληροφορίες που έχουμε, στις 10 Μαρτίου έλαβε μια ειδοποίηση από τον συνεισαγγελία ο κ. Φωκόπους, γιατί υποτίθεται ότι, δεν, ότι εργαζόταν χωρίς ε, ειδική άδεια ε, ως ανταποκριτής της Γκαζέτα Βιμπόσκα. η προειδοποίηση εξέπνευσε στις 23 Φεβρουαρίου 2009, δεν παρατάθηκε η άδειά του, ενώ τα άρθρα του συνέχισαν να εμφανίζονται στο site της εφημερίδας. Και πάλι κρατήθηκε στις 6 Απριλίου στη Χότνα ο κ. Βοσκόποτη γιατί παραβίασε τις συνθήκες ε, ε, υπό όρους απελευθέρωσής του και ήταν... Ε, ε, ε, και παρακολούθησε μία βιντεοσυνεδρίαση για τις αντιπροσωπείες μάλλον θα παρακολουθούσε μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στο ΜΙΣ. Και έκτοτε ο κ. Ποσκόπου κρατείται σε προδικαστική ε, φυλάκιση στην ε, φυλακή 1 του Πρότνατ, σύμφωνα με τον συνεταίρο του κυρίου ...σε επιτράπηκε στη σύζυγό του να τον επισκεφθεί την 1η Μαΐου. Από ό,τι φαίνεται ο κ. Ποσκόπους είναι σε θέση να στέλνει και να λαμβάνει η ενώ δεν έχουν, έχουν γίνει λίγες και καθόλου ανακρίσεις. Επιπλέον στις 13 Μαΐου ο κ. Βοσκόμπουτ επισήμως κατηγορήθηκε για προσβολή του Προέδρου υπό το άρθρο 368 του ποινικού κώδικα και για δυσφήμιση του Προέδρου ε, σύμφωνα με το άρθρο 367. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν μέχρι δύο έτη ή και τέσσερα έτη κάθριξης. Ε, οι αρχές αδιάκοπτα πιέζουν τον κύριο Προσκόπους όσον αφορά, που φαίνεται να είναι αντίπεινα για τις δημοσιογραφικές του δραστηριότητες. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης Τομής και εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις για αυτή την υπόθεση αλλά και για άλλες παρόμοιες. Στις 10 Απριλίου ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ της εκπροσώπου Κάθη Άστον εξέδωσε δήλωση για την έφοδο στα ανεξάρτητα ΜΜΕ στη που έχει ως εξής. Εκπρόσωπο ε, για τι εξωτερικέ υποθέσει και την ε, πολιτική ασφάλεια ανησυχεί ιδιαίτερω για την κατάσταση του κ. Ποσκόπου, που είναι ανταποκριτή τη Κασέτα Βιμπόσκα τη Πολωνική Καθημερινή Εφημερίδα κατά τη διάρκεια αποστολή του στο Μίνσκ τη Λευκορωσία. Ακόμα ένα παράδειγμα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζονται από πλευρά των αρχών τη Λευκορωσία μετά από τι προεδρικέ εκλογέ το Δεκέμβριο του 2010. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στεναρά καταδικάζει κάθε παρενόχληση φυλάκιση ή ε, παρεμπόδιση των ανεξαρτήτων ΜΜΕ καθώς και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η ελευθεροτυπία, η ελευθερία των ΜΜΕ και η ελευθερία έκφρασης ε, στην χώρα. Καλεί την Λευκορωσία να πάψει την δίωξη των ε, ανθρώπων αυτών και καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να συνεργαστούν ε, στενά με τους εκπροσώπους της ΟΑΣΕ για την ε, ελευθεροτυπία. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει πρόσβαση σε όλα τα άτομα που κρατούνται ως πολιτικοί κρατούμενοι και έχει καταδικάσει τις διαρκείς παρενοχλήσεις στην αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία. Χρησιμοποιούμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς και την μόνιμη πολιτική πίεση για να στηρίξουμε τον κύριο Ποσκόπουζ αλλά και άλλα θύματα καταπίεσης στις προσπάθειές τους ε, να υπερβούν εξαιρετικά δύσκολη και ανησυχητική κατάσταση. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, αυτή είναι η απάντηση της ΥΠΑ της εκπροσώπου, την οποία διαβιβάσαμε στον κύριο Καμίνσκι και την οποία θα διαβιβάσω εκ νέου με συνοδευτική επιστολή του κυρίου Ποπόφσκι, που είναι μάλιστα στα πολωνικά. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ επισήμως ε, και από τον κύριο Καμίνσκι να είναι ικανοποιημένος από την απάντηση που έλαβε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, είμαι ικανοποιημένο με την απάντηση την οποία έλαβα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την απάντηση αυτή. Ε, είναι πολύ σημαντικά λόγια και θα ακουστούν και στη Λευκορωσία και στην Πολωνία. Σας βεβαιώ γι' αυτό. Η Πολωνία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα αυτό και αυτό επιβεβαιώνει απλά και μόνο την υψηλή εκτίμηση και που τρέφω για την είπατε εκπρόσωπο αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υπηρεσία αυτή δεν ξεχνά ότι αυτό το οποίο μας ενώνει πέραν των θεμελίων που είναι οι συνθήκες είναι μια κοινότητα αξιών και ένα στοιχείο, μια αξία είναι η ελευθερία ε, λόγου και η δημοκρατία. Είμαι υπερήφανος που η υπηρεσία εξωτερικής δράσης προσπίζεται ενεργά αυτές τις αξίες. Γι' αυτό θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, για να απευθύνω έκκληση σε εσάς. Πρέπει να παρακολουθείτε στενά. Ποιοι αξιωματούχοι του καθεστώς Λουκασέγκο ενεργά προβαίνουν σε ενέργειες ε, παρενόχλησης ε, και καταστολής ε, των μελών της αντιπολίτευσης και θα πρέπει σε αυτά τα άτομα να επιβληθεί παγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τέλος να εκφράσω την ελπίδα μου ότι όλες αυτές, όλα αυτά τα κολλήματα, τα διαδικαστικά, ε, θα λυθούν και ελπίζω όλοι να μάθουμε πώ θα εργαζόμαστε και θα λειτουργούμε στη νέα πραγματικότητα με τη Συνδίκη τη Λισαβόνα. Παρ' όλα αυτά, γενικώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Στο περιθώριο αυτή τη κατάσταση ίσω ε, θα άξιζε τον κόπο να σκεφτούμε πώ θα οργανώσουμε μια πιο γρήγορη και εύκολη ε, διαδικασία για την ώρα των ερωτήσεων, ώστε να έχουμε απαντήσεις από πλευρά του εκτελεστικού πιο παρκής και που θα ανταποκρίνονται στις ε, απαιτήσει των βουλευτών. Η ώρα των ερωτήσεων είναι μια διαδικασία που ισχύει σε διάφορες χώρες και μπορούμε να το αναπαράγουμε και εδώ, στο δικό μας κοινοβούλιο. Επόμενο σημείο είναι το 14. Ε, α, ανταλλαγή απόψεων, ε, μα, συγγνώμη, ο απολογισμός της επίσκεψης ε, στο Ιράκ στις 24 με 26 Απριλίου είναι μια έκτακτη επίσκεψη. Ε, πρώτη φορά γίνεται γιατί παλιότερα τους, δεν, δεν υπήρχε πρόσβαση στο Ιράκ για λόγους ασφαλείας. Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τους κυρίους Στίβενσον, Μάουρο, Μολτάντιν και Κάλτσιν και επισκέφθηκαν τη Βαγδάτη και την Έρβιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε πολύ σωστά. Ήταν μοναδική αυτή η περίπτωση γιατί τη δημιουργήσαμε ως επίσημη αντιπροσωπεία αυτή μετά, μόλις μετά τις τελευταίες εκλογές. Δυο φορές πριν μας αρνήθηκαν ε, την είσοδο στο Ιράκ για λόγους ασφαλείας. Η δική μας η διάσκεψη των Προέδρων αρνήθηκε. Διαμαρτυρηθήκαμε λοιπόν και με τη βοήθεια της Επιτροπής αυτής αλλά και με τη βοήθεια των Προέδρων των Αντιπροσωπιών, της διάσκεψης Προέδρων Αντιπροσωπιών πήραμε τελικά την έγκριση. Πρέπει να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης είδαμε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη το μόνο πρόσωπο που δεν είδαμε ήταν ο Πρωθυπουργό Νουριά Μαλική που ήταν τότε στη Νότιο Κορέα. Αλλά είχαμε το προνόμιο να δούμε τον πρόεδρο Ταλαμπανή, τον πρόεδρο του Ιράκ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο Σάμαν Τζέιφι, το Συμβούλιο Αντιπροσώπων που είναι το μόνο τμήμα της κυβέρνησης που λειτουργεί, θα το αναφέρω και μετά αυτό, είδαμε τρεις επιτροπές από το Κοινοβούλιο, ασφάλεια άμυνας, εξωτερικών υποθέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είδαμε τον ε, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μούτλακ, ο Υπουργός Εξωτερικών Σαμπαρή, ε, ήρθε μαζί με τον εκπρόσωπο του Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ε, μάλιστα μετά από πρόσκληση πρόσφατα ήρθε και επισκέφθηκε τη δική σας επιτροπή. Είχαμε συναντήσεις με τον Αμερικανό πρεσβευτή Jim Jeffrey με την ΕΕΔ ε, προφανώς για να κανονίσουμε το πρόγραμμα και μας συνόδευε και ο Πολωνός πρεσβευτής στο Ιράκ ο Στάνισλαβ Σμόλεν ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. Στην Ερμπίλ είδαμε τον πρόεδρο Μασούτ Μπαρζάνη πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν τον πρόεδρο του Κουρδικού Κοινοβουλίου Καμάλ Κακούκη, τον πρωθυπουργό Δόκτωρα Μπάρεμ Σάλε. Επίσης συναντήσαμε και τον επικεφαλής της ε, Ρακία, τον Δόκτωρα Λάουι, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στην Ερμπίλ εκείνη την εποχή, και τον κυβερνήτη της Ερμπίλ, τον Νόβατ Χάντι, τον επίσκοπο Μπάσαρ Μάρτι Βόρντα, στο, από την Ερμπίλ για να δούμε τα προβλήματα της χριστιανικής μειονότητας και ε, ηγέτες του κόμματος της αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν. Τα βασικά θέματα ήταν η Αραβική Άνοιξη, που εξετάζεται με μεγάλη σοβαρότητα, ακόμα και πιο, με μεγαλύτερη ένταση συζητείται το θέμα από εκείνους, από ό,τι ίσως και από, εδώ από εμά γιατί το θεωρούν αυτό ισοδύναμο της πτώσης του τείχους του Βερολίνου. Υπάρχουν φόβοι όμως ότι για παράδειγμα στη Συρία όπου υπάρχει πολύ μεγάλη κουρδική κοινότητα και πολλοί χριστιανοί ότι μπορούν να φύγουν από τη βία στην Συρία και να πάνε στο Κουρδιστάν για ασφάλεια. Το Κουρδιστάν, μας είπαν επανειλημμένα, κατακλείζεται ήδη από πρόσφυγες ποτέ δεν διώχνουν κανένα, αλλά έχουν έλλειψη στέγη, σχολείων, κλινικών, νοσοκομείων. Και μάλιστα ο Επίσκοπος ε, Μπόρντα μας είπε ότι μας παρακαλεί να ενημερώσουμε τους συναδέλφους στην Ευρώπη να μην στέλνουν ε, οικονομικούς πόρους στο Κουρδιστάν για να οικοδομούν καινούργιες χριστιανικέ εκκλησίες. Θέλουμε νοσοκομεία, κλινικές, σχολεία, σπίτια, όχι εκκλησίες, για τους εκτοπισμένους χριστιανούς, εκ των οποίων δεκάδες χιλιάδες αναζήτησαν ασφάλεια στο Κουρδιστάν. Συζητήσαμε όλη την πολιτική κατάσταση στο Ιράκ βεβαίω, Η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας που ανέλαβε 8 μήνες μετά τις ε, περσινές εκλογές για να σχηματίσει επιτέλους μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας που είναι γνωστή ως η συμφωνία της Ερμπίλ με νέα ρήτρες που συνδυάζουν τα διαφορετικά, ε, τις διαφορετικές συνιστώσεις της του μεγάλου συνασπισμού. Καμία από τις εννέα ρήτρες της συμφωνίας της Ερμπίλ δεν έχει εφαρμοστεί, ούτε μία. Τα τρία κύρια Υπουργεία, Υπουργείο Ασφάλειας, Άμυνας και Εσωτερικών, που είναι κέρια σημασίας και αποτελούν τμήμα της Συμφωνίας Ερμπίλ γιατί θα έπρεπε να δοθούν σε κάποια από τα συμμετέχοντα κόμματα του συνασπισμού δεν ε, ορίστηκαν ποτέ και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των Υπουργών βρίσκονται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Έτσι ο Πρωθυπουργό ε, Νουριά Μαλική έχει τεράστιες ευθύνες και μεγάλη εξουσία στο Ιράκ. Επίσης, ε, το Εθνικό Συμβούλιο Στρατηγικών Πολιτικών που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να συγκροτηθεί υπό την ηγεσία του Χάρια Αντάλουι από το κόμμα Αγιαρακία που ε, έχει μία έδρα παραπάνω από το κόμμα Ντάουερ του Μαλική στις εκλογές αν και ο Νούρια Μαλική τελικά έγινε πρωθυπουργό. Αυτό το Εθνικό Συμβούλιο λοιπόν Στρατηγικών Πολιτικών ε, δεν συγκροτήθηκε, παρόλο που προβλέπεται από τη Συμφωνία της Ερμπίλ. Πολλοί πολιτικοί ηγέτες, ε, συνομιλητές μας, είπαν ότι προβλέπουν πάλι πρόορες εκλογές. Γιατί υπάρχει πραγματικά συμφόρηση στην κυβέρνηση τώρα. Ε, ένα από τα λίγα νομοσχέδια που πέρασε από τη Βουλή ε, ήταν για τον προϋπολογισμό. Πολλά άλλα νομοσχέδια κόλλησαν και δεν προχωρούν γιατί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας δεν λειτουργεί κανονικά. Παρόλα αυτά, μιλήσαμε για την οικονομική κατάσταση, λόγω της κατάστασης ασφαλείας που είναι ακόμα προβληματική στη Βαγδάτη και το είδαμε με τα μάτια μας. Είδαμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ακόμα η πόλη. 81 ε, αστυνομικοί ε, δολοφονήθηκαν τις 16 μέρες πριν πάμε εμείς. Αυτά τα πράγματα εμείς σπάνια τα ακούμε εδώ. Μας έδειξαν ε, σημεία ε, ε, μεγάλων οπών ε, από βόμβες κοντά στα σημεία ελέγχου που σκότωσαν πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πλήγματα, επιθέσεις, δολοφονίες. Είναι στην ημερήσια διάταξη ακόμα στη χώρα. Υπάρχει περιορισμένη ηλεκτροδότηση σε περιοχές όπως η Βαγδάτη, στη, στη Βαγδάτη. Πολλές φορές κόβεται για έξι ώρες ε, το ηλεκτρικό. Αργότερα το, με το Ραμαντάν και που θα ανέβει στη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς και η μουσουλμανική κοινότητα δεν θα μπορεί ούτε να τρώει ούτε να πίνει τις ε, ώρες της ημέρας, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όλα αυτά γίνονται πολύ επικίνδυνα όταν δεν υπάρχει ε, ηλεκτρικό και δεν υπάρχει κλιματισμός. Και μπορεί να αυξηθούν τα κρούσματα βίας μετά από αυτά, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Ε, υπάρχει αύξηση παραγωγής πετρελαίου και αερίου και γιατί θέλουν να δώσουν ε, έναυσμα στην οικονομία και στο Κουρδιστάν είδαμε εμείς πώς έχουν αιτήσει αύξηση κάθε χρόνο 10%. Το Κουρδιστάν ανθεί οικονομικά γιατί η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια εκεί είναι πολύ καλύτερη. Δηλαδή είναι αρκετά ασφαλές τμήμα του Ιράκ, του Κουρδιστάν. Ένα από τα κέρια ζητήματα βέβαια που εθέσαμε εμείς σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε ήταν η σοβαρή μας ανησυχία και σοβαρή μας διαμαρτυρία για το λουτρό αίματο στο Καμπάσεφ στις 8 Απριλίου φέτος όπου ε, δολοφονήθηκαν 35 άμαχοι, άοπλοι. Ε, δολοφονήθηκαν από τις δυνάμεις του Ιράκ και πολλοί τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Ε, η πολιορκία συνεχίζεται, ε, φαρμακευτική περίθαλψη και ιατρική περίθαλψη δεν παρεσχέθη όπως έπρεπε στους τραυματίες και ο Αλ Μέρκετ από το Δυνάμι είπε στην αντιπροσωπεία μας ότι η μόνη πιθανή λύση είναι να φύγουν οι 3.400 από το Ασράφ έξω από το Ιράκ. Πρέπει όμως, ε, μας είπαν, να πιστεί η ηγεσία του MK που είναι η Μουτζαχεντίν του λαού. Πρέπει οι ηγέτες των Μουτζαχεντίν, όχι μόνο στο καταβλισμό Ασράφα, αλλά και στο Πάρες ότι αυτή είναι η λύση. Όταν γύρισα από το Ιράκ, αμέσως φρόντισα να πάω στο Πάιρος. Πήγα και μίλησα με τους ηγέτες του MK πέντε ώρες στο Πάιρας και τους έπεισα να συμφωνήσουν σε μια εναλλακτική που συμφωνήθηκε α, μεταξύ αντιπροσωπείας μας, από την αντιπροσωπεία μας για το Ιράκ και πάνω σε αυτό έγινε και μια συνέντευξη τύπου στο Στρασβούργο στην προηγούμενη Ολομέλεια στα άλλη στη Βαρόνια Άστον και στους ε, υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών, 27. Η επιλογή είναι η επανεγκατάσταση των 3.400 κατοίκων του στο Άστραφ σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη-μέλη όπου έχουν μέλη της οικογένειας, κάποιους, κάποια διασύνδεση και στις ΗΠΑ, Καναδά, Νορβηγία, Ελβετία, Αυστραλία, όποια χώρα που μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα και να αποφύγουμε περαιτέρω σφαγή και ε, Γιατί οι Ιρακινοί το ξεκαθάρισαν. Θέλουν να λυθεί μέχρι το τέλος του χρόνου το πρόβλημα αυτό. Όμως ε, θέσαμε έναν αυστηρό όρο μετά από συζητήσεις ε, με τους ε, πρέσβεις των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ. Είπαν ότι δεν μπορούμε να θεωρηθεί, δεν μπορούμε να Ανταμείψομαι σε εισαγωγικά για τη σφαγή του Ιρακινού, απομακρύνοντας όλον αυτόν τον κόσμο από το Ιράκ που αυτό ακριβώς θέλαν ούτως ή άλλως οι Ιρακινέ αρχέ. Η λοιπόν, άλλω οι ιρακινέ αρχες η προυποθεση λοιπον που εθεσαμε με αρχές θα πρέπει να αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις ε, κατοχής στον καταβλισμό Ασράφ, πρέπει να τεθεί τέλος στην πολιορκία να επιτραπεί στους δημοσιογράφους και τους ανεξάρτητους παρατηρητές να εισέλθουν στον καταβλισμό, να παράσχουν ε, κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους σοβαρά τραυματίες και να καλέσουν μια ε, διεθνή έρευνα ε, που θα εξετάσει τη σφαγή τα, τα, τα γεγονότα της 8ης Απριλίου. αν δεχθούν τους όρους θα καταλάβουμε ότι θα θελήσουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση. Το Άσραφ ήταν στην ατζέντα των Υπουργών Εξωτερικών της Δευτέρας αυτή τη βδομάδα όταν η Βαρόνι Άστον έθεσε το θέμα και διαμαρτυρήθηκε και πάλι στην Ιρακινή κυβέρνηση για τη σφαγή. Οπότε κινούνται τα πράγματα ως προς το θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη που χρειάζεται για να επιληθεί το πρόβλημα και να μην γίνουμε μάρτυρες κι άλλης φαγής. Επίσης προτείναμε να γίνει μια διάσκεψη για, με, για επενδύσεις το Δεκέμβριο φέτος, 6 και 7 Δεκεμβρίου, μαζί με την Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να εξετάσουμε την παραγωγή, την πιθανή πετρελαίου αερίου και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις στη χώρα. Να δούμε και τον τομέα της γεωργίας τις ε, δημοσιονομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Κομισιόν το είδε με ενθουσιασμό το θέμα και η Πολωνική Προεδρία ήδη υποσχέθηκε ότι αυτό το θέμα θα το αναδείξει ε, ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της ως κύριο θέμα. Οπότε ήταν χρήσιμη αυτή η πρωτοβουλία μετά από την επίσκεψή μας. Επίσης, υπογράψαμε την κοινή διακήρυξη η οποία ζητεί να εφαρμοστεί το, η συμφωνία συνεργασίας που υπογράφει πέρσι και ζητούμε εταιρική σχέση, συμπράξει περισσότερε σε θέματα κοινωνικά, ανθρώπινα δικαιώματα, παιδεία, θέματα ισότητα των φύλων, προβλήματα των γυναικών. Οπότε γενικά ήταν μια πολύ χρησιμότατη σειρά συναντήσεων αυτή και προσβλέπουμε στο μέλλον να καλωσορίσουμε κάποιους από τους Ιρακινούς που συναντήσαμε στην Ευρώπη, μάλιστα η Υπουργή, ο Υπουργό Ενέργειας θα έρθει αυτή τη βδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, για να συναντήσει τον Επίτροπο Ότιμιρ. Οπότε περιμένω ότι θα έχουμε επικοδομητική συνεργασία με τους Ιρακινούς στο μέλλον. Να πω τέλος κύριε Πρόεδρε ότι είμαι πολύ ευγνώμων στην Επιτροπή αυτή που μου έδωσε τη δυνατότητα να έρθω για να μιλήσω σήμερα. Επίσης ε, λυπάμαι διότι μου είπατε ότι συμμετείχα και ήμουν συμπρόεδρος σε μια συνεδρίαση για κοινωνικά θέματα για το Ιράκ σήμερα το απόγευμα. Αλλά ε, αυτό έγινε χωρίς να ενημερωθώ και ήδη προεδρεύω σε μια άλλη συνεδρίαση για το Ιράκ σήμερα το απόγευμα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην ε, καινούργια αυτή συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε για αυτό. Εγώ το γνώριζα. Ήξερα πώς έχει κατάσταση. Οπότε θα προσαρμοστούμε για το μεσημέρι. Ο κύριος Μάρο τώρα θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη είπε ο συνάδελφος Στίβενσον. Γι' αυτό περιορίζομαι να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τα όσα εκείνος δεν ανέφερε και φαντάζομαι ότι θα τα επαναλάβουμε και στην απόψενή ακρόαση. Το παράδοξο είναι ότι στο Ιράκ πεθαίνει ε, κανείς ε, επειδή θέλει να ζήσει. Πεθαίνουν δηλαδή αυτοί που δεν εγκαταλείπουν ε, την προσπάθεια. Συνεχίζουν να πηγαίνουν να δουλεύουν, συνεχίζουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στον εκδημοκρατισμό της χώρας. Και είναι αντιφατική και η θέση των δικών μας θεσμικών οργάνων σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο Ιράκ. Να σας δώσω παραδείγματα τα οποία ήδη έχω δώσει στη συζήτηση που κάναμε με την ε, κυρία Άστον στη κοινή συζήτηση στην Ολομέλεια. Δηλαδή διαπιστώσαμε την απόλυτη ανεπάρκεια της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιπροσωπεύει στο Ιράκ. Δηλαδή, εξηγούμε, τα άτομα μεμονωμένα είναι με μεγάλ, έχουν μεγάλα προσόντα, είναι αφοσιωμένα και είναι και επικεντρωμένα στην εργασία τους. Αλλά μιλάμε για δύο ανθρώπους όπου τώρα θα προσθεθεί και η πρέσβης η Μπασκόβα που ενεργούν μέσα στο βρετανικό θύλακα, δηλαδή στην ουσία δίνουν μια εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτάται απόλυτα από πλευράς μιας εκ των δυνάμεων που τα τελευταία χρόνια ενήργησαν στο Ιράκ για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και με την άφηξη της κυρίας Συμπασκόβα πρόκειται για τρεις ανθρώπους. Και για να εξηγήσω πόσο ανεπαρκής είναι αυτή η κατάσταση, ε, ε, ε, υπογράμμισα ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Μπαχάμες βασίζεται σε 7 υπαλλήλου. Εγώ δεν θέλω να κάνω λαϊκιστικού τύπου δηλώσεις και ενέργειες, αλλά Α συνειδητοποιήσουμε ότι μια χώρα με 40 εκατομμύρια ανθρώπου που έχει στρατηγική και ιστορική και πολιτιστική και πολιτική σημασία όπω το Ιράκ και που άρα θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει για την Ευρώπη Εκείνη την Ευρώπη που διχάστηκε τη φάση του πολέμου θα έπρεπε να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για να δώσουμε μια εικόνα κοινή εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτή τη φάση σίγουρα ε, χαίρει μιας παρέμβασης πολύ κατώτερης ε, σε σχέση με την, τη σημασία των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και η δεύτερη μου παρατήρηση ε, αφορά το στρατόπεδο Ασράφ. Να προσθέσω στα όσα είπε ο Στρούαν Στίβενσον ότι οι πληροφορίες που έχουμε για επιστροφή του Συμβουλίου από το... Μάλλον τα όσα ακούσαμε από το Συμβούλιο των Υπουργών της Δευτέρας δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Δηλαδή ένα πρόβλημα τέτοιου τύπου θα, λυθεί στην περιφέρεια. Μα η ανθρωπιστική κατάσταση στο στρατόπεδο Ασράφ θα λυθεί στην περιοχή, θα πει ότι είτε λύνει το πρόβλημα το Ιράκ είτε το Ιράν. Είτε ο ένα είτε ο άλλο είναι ακατάλληλο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, συνειδητά, αυτή τη στιγμή, ελπίζω πως αύριο μεθαύριο δεν θα παραστήσει κανεί ότι δεν άκουσε και δεν είδε τι γίνεται. Εμείς στην ουσία συνειδητά εκθέτουμε αυτού του 3.000 ανθρώπου σε έναν σοβαρό κίνδυνο γιατί δεν έχουμε τη θέληση να αναλάβουμε ευθύνες συγκεκριμένες σε σχέση με την μοίρα τους. Και μιλώ προφανώς από ανθρωπιστικής άποψης και μόνο. Δεν θέλω να μιλήσω για να κάνω αξιολογήσεις πολιτικής φύσης ε, που θα ήταν περίπλοκες και των οποίων την περιπλοκότητα είδαμε και επί Διότι το όσο στο Ιρακινό Κοινοβούλιο όσο και στις επαφές με τον Αμερικανό πρέσβη, πρέσβη οι πολιτικής φύσης δυσκολίες που κρύβονται πίσω από το στρατόπεδο Ασράφ είναι πολύ μεγάλες. Επόμενη παρατηρήσή μου αφορά το θέμα των μειονοτήτων που προφανώς σε ένα που έχει, σε μια περιοχή μάλλον που έχει πρόβλημα σταθεροποίηση είναι πολύ σημαντικό. Ως προς αυτό λοιπόν να παραθέτω την ε, επαφή που είχαμε με τον πρόεδρο Στίβενσον και τους υπόλοιπους συναδέλφους στην Ερβίλ με τον ε, καθολικό αρχιεπίσκοπο Καλντέο που μας έθεσε ενώπιον μιας ψυχής και έπειτα ε, έκανε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο Παρζάνη ε, Μα έθεσε ενώπιον λοιπόν μια πολύ σημαντική κατάσταση. Μέχρι στιγμή μιλούσαμε για του χριστιανού που φεύγαν από το Ιράκ, ξέφευγαν προ τη Συρία και στην Ιορδανία. Προσοχή όμω γιατί τα όσα συμβαίνουν στη Συρία μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πρόβλημα όσον αφορά την επιστροφή αυτών των ανθρώπων ε, την επιστροφή την ε, βιαστική λόγω των σοβαρών ε, γεγονότων στη Συρία θα μπορούσαμε λοιπόν να βρεθούμε ενώπιον ενός νέου κεφαλαίου ανθρωπιστικής επίγουσας ανάγκης που μπορεί να επιβεβαιωθεί στο Ιρακινό Κουρδιστάν που φαίνεται ότι είναι η μόνη περιοχή με βάση την καλύτερη κατάσταση που επικρατεί εκεί είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν σημαντικό στην συζήτηση με τους Κούρδους εθήνοντες ότι έπρεπε να θέσουμε στόχο ε, μια πιο σημαντική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερμπίλ. Δηλαδή να ε, υπάρξει εκεί μια ευρωπαϊκή εκπροσώπηση ε, ώστε να μπορέσουμε πιο εύκολα και πιο λειτουργικά να αναλάβουμε ευθύνες σε αυτή την περιοχή. Τελευταία παρατήρηση που έχω να προσθέσω σχετίζεται με τις επαφές στη Βαγδάτη και στην πολιτική σύγχυση που επικρατεί και που οφείλεται και στην κυβέρνηση Μαλίκη. Η πολιτική αναποφασιστικότητα επιδεινώνει με το πρόβλημα της ασφάλειας. Ε, αν δεν υπάρχει βούληση για υλοποίηση μιας ε, αυθεντικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, εφόσον το, αυτό είναι το αποτέλεσμα της κάλπης, ε, φυσικά η αστάθεια προκαλεί ανασφάλεια και με τη σειρά της ανασφάλεια προκαλεί και πολιτική αστάθεια. Άρα λοιπόν είναι, αναμένεται και είναι και σημαντική η φωνή της Ευρώπης και για αυτό το θέμα και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω έκκληση στο τέλος ε, αυτής της ε, αξιολόγησης της, ε, του ταξιδιού μας στο Ιράκ. Θέλω λοιπόν να το υπογραμμίσω τη σημασία της παρουσίας της, ε, της εκπροσώπου Άστον όσο γίνεται πιο σύντομα στο Ιράκ και κυρίως με προτάσεις που να μπορούν να παρουσιάζουν καταλήλως τη στρατηγική και τις λύσεις που μπορεί να προτείνει η Ευρώπη υπό αυτές τις συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως και θα ενημερώσουμε την είπατε εκπρόσωπο. Με βάση τα όσα μας είπατε. Και τώρα ο κύριος Τάνοκ και μετά ο κύριος Κέλλαν. Για να είμαι ειλικρινής κύριε Πρόεδρε, πολύ εύγλωτα με κάλυψε ο συνάδελφος Στίβενσον και ο συνάδελφος Μάουρο. Όλα όσα είχαν να πω έχουν διποθεί. Πράγματι υπάρχει ανεπαρκές προσωπικό, ανεπαρκείς πόροι που είναι διαθέσιμη ε, στην πρέσβη Γιάννα Ιμπάσκοβα που ήταν και τέος συνάδελφος. Πολύ μικρό, το, πολύ ολιγάριθμο το προσωπικό που έχει να αντιμετωπίσει τόσα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας δικαιωμάτων των μειονοτήτων, στο Ιράκ. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση σε εσά να μεταφέρετε την ανησυχία μα στην είπατε εκπρόσωπο και στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Σίγουρα έχουμε θέματα με το προπλησμό, δεν θέλουμε άξιο προπλησμό, αλλά το Ιράκ είναι προτεραιότητα. Όταν το προσωπικό τη κυρία ε, Μπάσκοβα είναι τέσσερα μόλι άτομα, καταλαβαίνετε ότι είναι ανεπαρκέστατο. Ευχαριστώ κύριο Σκέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Στίβενσον που κατέληξε σε μια πολύ ρεαλιστική λύση για αυτή την ε, μακροχρόνια ανθρώπινη τραγωδία στο στρατόπεδο Ασράφ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει και θα μπορούσε να δοθεί και ως μια μελέτη περίπτωσης, ε, ως ένα stress test για να δούμε ε, αν μπορεί να σεβαστεί τη δημοκρατική ανθρώπινα δικαιώματα το Ιράκ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη το ότι οι διαμένοντες σε αυτό το στρατόπεδο έχουν αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις γειτονίας ε, με τον πληθυσμό. Μαθαίνουν αραβικά, και πραγματικά στηρίζονται, τους στηρίζουν ενεργά οι γείτονές τους. Δεν είναι κάτι ε, ξένο δεν είναι ένα ξένο σώμα στο Ιράκ. Από τον Απρίλιο του 2009 έγιναν δύο επίσημες προσπάθειες ε, στήριξης από πλευράς Κοινοβουλίου, στήριξης της ακαιρότητας και των ζωών ε, της ε, αντιπολίτευσης, των μελών της αντιπολίτευσης. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι η Βαρόνια Άστον πλέον εκθέτει την κατάσταση, παζέζει αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε εκφραστεί πολύ νωρίτερα. Οπότε θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτή την τραγωδία. Επίσης, συμμερίζομαι τις ανησυχίες του συναδέλφου Μάουρο για άλλες μειονότητες, όπως είναι οι χριστιανοί στο Κουρδιστάν. Το τελευταίο σημείο που θέλω να φέρω είναι ότι στηρίζω πλήρως την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο Ιράκ που πραγματικά έχει τεράστιο δυναμικό. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ένας παράγοντας ε, σημαντικός στο παγκόσμιο προσκήνιο, πιστεύω ότι απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση και συγκέντρωση σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει επίσης σαφής ανάγκη εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να καταστεί δυνατή και στο Βόρειο Ιράκ, ε, στην Ερμπίλ για παράδειγμα. Thank you. Mr. Stevenson, please. Ευχαριστώ κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Να συμφωνήσω όλους ιδιαίτερως με τα σχόλια του Μάριο Μάουρο η συμμετοχή στην αντιπροσωπεία, εκ μέρους, η συμμετοχή του στην αντιπροσωπεία εκ μέρους της Επιτροπής ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και χρήσιμη. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπαν ε, ο Κέλαμ και ο Τάνοκ για την ε, ανεπαρκή παρουσία, ε, το ανεπαρκές προσωπικό της γιατί ΕΕ, αυτό είναι σαφές και μας το λένε και μας το ξαναλένε πρέπει, είναι σημαντικό να επισκέπτεται το Ιράκ η κάθε άστο. Δεν έχει, ε, έχει πάει σε άλλες χώρες περιοχής, αλλά πρέπει να μεταβεί στο Ιράκ για να δει πόσο ανεπαρκές το προσωπικό της υπηρεσίας στη χώρα αυτή. Και πρέπει να αναβαθμιστεί η παρουσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο στράπετα ο Αμερικανό πρέσβης, ουσιαστικά θόλωσε τα νερά με μια πρόταση που διατύπωσε για μετακίνηση των 3.400 ατόμων που είναι στο Ασράφ σε μια πρώην Αμερικανική στρατιωτική βάση. Τα άτομα αυτά, τα άτομα που είναι στο Ασράφ, αρνήθηκαν εντελώς. Είπαν αν να πεθάνουμε ε, στο Ιράκ, ας πεθάνουμε στην Ασράφ και δεν χρειάζεται να πάμε κάπου αλλού για να πεθάνουμε. Ε, το Ιράν το οποίο πίεζε την αποξένωση ε, αυτού του στρατοπέδου και ασκούσε πίεση στην Ιρακινή κυβέρνηση το γεγονός ότι έχουν απορρίψει οι ίδιοι την εκτόπιση, τη μετακίνηση αυτών των 3.400 ατόμων εκτός Ιράκ δείχνει ότι μάλλον δέχονται την ε, αμερικανική επιλογή μετατόπισης τους εντός Ιράκ. Και αυτό ε, πραγματικά είναι μια επικίνδυνη επιλογή. Θα οδηγήσει σε σφαγές ε, είδους τύπου Σρεμπρένιτσα. Θα πρέπει αυτή η ιδέα να μην ευδοκιμήσει. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη λύση που έχουμε προτείνει εμείς και την οποία οι ίδιοι οι διαμένοντες εκεί φαίνεται να τη στηρίζουν. Ευχαριστώ. Thank you um, Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 3 θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Έχουμε μια κράση για τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις στο Ιράκ. Θα επακολουθήσει παρουσίαση από τον Επιτρόπο Φίλε. Παρουσίαση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Αλλά θα μας ε, εκθέσει και την σχεδόν οριστικοποιημένη άποψή του για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Ελπίζω να σας δω στις τρεις και όχι μόνο εσάς, να δω και πολύ περισσότερους. Ευχαριστώ.